Μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Θα σας θυμίσω, όπως ε, και τις άλλες φορές, ότι αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται από την υπηρεσία ίντερνετ. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω τον κύριο Λούκαση εδώ στο Προεδρείο και το νέο μας διοικητικό υπάλληλο στην ε, Γραμματεία που είναι ο κύριος που είναι Ουγγαρέζος και έχει ήδη δουλέψει σε διάφορες επιτροπές αλλά όχι σε τούτη. Του ευχόμαστε λοιπόν ε, να εργαστεί ικανοποιητικά στην ε, συνεδρίασή μας ε, και χαιρόμαστε για τη γνωριμία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα πρέπει να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Η σημερινή συνεδρίαση θα γίνει μόνο το σήμερα το απόγευμα γιατί αύριο όπως είναι γνωστό υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν τη νέα επιτροπή και άρα είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε. Μόνο απόψε λοιπόν θα συνεδριάσουμε. Μετά από τη συνεδρίαση θα γίνει η συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε να θυμίσω στους συντονίστες ότι θα πρέπει να μείνουν λίγο παραπάνω μετά το τέλος της συνεδρίασης. Η ημερήσια διάταξη σας έχει ήδη διανεμηθεί, θα την έχετε διαβάσει πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο συνάδελφο Ράγκελ ζήτησε να ε, βάλουμε στην ημερήσια διάταξη μια ανταλλαγή απόψεων για τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε καμία δυσκολία να το κάνουμε. Να ρωτήσω αν υπάρχουν δυσκολίες, δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Οπότε το ε, εντάσσουμε στην ημερήσια διάταξη και Φαντάζομαι ότι εγκρίνεται και την υπόλοιπη μερίσια διάταξη από τις οποίες το συμπεραίνω. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Ράγκελ για την συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω ότι έχουμε διοργανώσει διάφορες συνεδριάσεις, αρκετές. Καταρχήν μόνο μεταξύ των διαφόρων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους έξι που συναποτελούν την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως γνωρίζετε, ηγείται αυτής ο κύριος Λένε. Ο κύριος Λένε είχε μία συνεδρίαση με τον πρόεδρο Μπαρόζο όπου αποφάσισαν οι δυο τους το πλαίσιο της συμφωνίας πλαισίου και στη συνέχεια είχαμε δύο συνεδριάσεις με τον πρόεδρο Παρόζο, πολύ καρποφόρες. Αύριο έχουμε μια πολύ πολύ σημαντική συνεδρίαση ανάμεσα στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αντιπροσωπεία της Κοπισιόν όπου θα προεδρεύσει ο κύριος Λένε από πλευράς Κοινοβουλίου και ο κύριος Μπαρόζο από πλευράς Κομισιόν. Θα συμμετέχουμε όλοι σε αυτή τη συνεδρίαση. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε επιτύχει μερικά πράγματα. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί όπως γνωρίζετε ε, υπάρχουν κάποια εμπιστευτικά στοιχεία σε σχέση με αυτό το ζήτημα αλλά θα έλεγα ότι Έχουμε επιτύχει κάποιες από τις ε, προϋποθέσεις μας σε σχέση ε, με το θέμα της πρωτοβουλίας, επίσης με το θέμα με το θέμα της ψήφου μομφής προς έναν ε, συγκεκριμένο επίτροπο επίσης τις διεθνείς σχέσεις, επίσης για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα πρέπει οι επίτροποι να συμμετέχουν ε, και στις συζητήσεις στην ε, Ολομέλη και εδώ έχουμε επιτύχει κάποια πράγματα. Να σας πω επίσης ότι όλα αυτά είναι συμβατά και σύμμορφα με την συνθήκη της Λισαβόνας κάποιες φορές την ξεπερνούν κάπως, αλλά όχι, δεν είναι εναντίον της. Και όταν ξεπερνούν την διατυπώσεις της συνθήκης Λισαβόνα, συνήθως ε, αντιπροσωπεύουν ε, και κέρδος για το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η κατάσταση πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω πως είναι μια πολύ λογική συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις ε, βρίσκονται σε πολύ καλή φάση. Οι σχέσεις έχουν διευκολυνθεί γιατί και τα δύο μέρη δέχονται ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει κάποιες ε, νέες ε, αρμοδιότητες και δέχονται πως υπάρχουν όρια στην συνθήκη της Λισαβόνας σε σχέση με αυτές τις ε, αρμοδιότητες. και θα έλεγα πως έχει βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο θέσεις και πιστεύω πως μπορούμε να έχουμε τις βασικές κατευθύνσεις γραμμές της Συμφωνίας Πλαισίου ίσως και αύριο ή και μέσα στην εβδομάδα αυτή. Βεβαίως πρόκειται μόνο για πολιτική φύσης κατευθύνσεις γραμμές, είναι μόνο τα σπουδαιότερα σημεία, αλλά για μάς είναι πολύ σημαντικό να συναυθεί αυτή η συμφωνία πριν να ψηφιστεί η Κομισιόν. Αυτός είναι ο στόχος μας. Βέβαια, οι τεχνικές πτυχές θα αναπτυχθούν μετά από την ψήφο για την Επιτροπή και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί πλήρω η συμφωνία μόνο γύρω στο Πάσχα. Είμαι λίγο μετά το Πάσχα. Πάντω, τα πολιτικά επιτεύγματα του Κοινοβουλίου σε σχέση με την Κομισιόν, αυτές, ε, αυτά τα επιτεύγματα, αυτέ οι ε, νέε αρμοδιότητε που προσπαθούμε να κερδίσουμε θα έχουν κλείσει και αποφασιστεί πριν από την ψηφοφορία για την Κομισιόν. Εντύπωσή μου είναι λοιπόν ότι, ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την συνένεση ανάμεσα στις διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες τους ε, εκπροσώπους των φιλελευθέρων, των πρασίνων, των σοσιαλιστών και του ΕΛΚΑ και η στάση που έχει αναπτύξει η Κομισιόν μετά από κάποια αρχικές ε, διαπραγματεύσεις που ήταν κάπως τεταμένες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερες εξελίξεις στις θεσμικές σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν και λιγότερες εξελίξεις σε τομείς όπως για παράδειγμα οι διεθνείς σχέσεις. Κάτι το οποίο δεν ήταν βέβαιο και που τώρα πλέον είναι δεδομένο είναι η συμμεταχείριση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από πλευρά τη Κομισιόν. Η Κομισιόν αναγνωρίζει λοιπόν πω μετά από τη συνθήκη τη Λισαβόνα θα έχουμε το ίδιο είδος ενημέρωσης και το ίδιο χρονοδιάγραμμα ώστε να λαμβάνουμε τις πληροφορίες και την ενημέρωση ταυτόχρονα με το Συμβούλιο. Και αυτό είναι μεγάλο η επιτυχία όσον αφορά την επικοινωνία και την ενημέρωση από πλευράς της Κομισιόν που έχει την πρωτοβουλία και των δύο νομοθετικών σωμάτων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Είναι πλέον ένα ισοσκελές τρίγωνο, είμαστε σε, στην ίδια θέση με το Συμβούλιο. Αυτή είναι η ουσία λοιπόν των διαπραγματεύσεων και πιθανότητα μεθαύριο, αύριο μεθαύριο θα έχουμε περαιτέρω ενημέρωση. Φυσικά θα τα πω πρώτα στη, στη διάσκεψη των Προέδρων και μετά στην Επιτροπή μας που είναι η αρμόδια για να α, ενημερωθεί για τη Συμφωνία Πλαίσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που κάνατε, για τις προφορίες που μας δώσατε. Αν κάποιο τώρα θέλει να πάρει το λόγο για αυτό το σημείο, έχει το λόγο. Αν δεν βλέπω κανένα υψωμένο χέρι. Ευχαριστώ τον κύριο Ράγκελ για τις πληροφορίες. Και χαιρόμαστε και το εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την γρήγορη εξέλιξη σε αυτό το σημείο. Πάμε στο δεύτερο σημείο, ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το ΕΛΚ διόρισε τον κύριο Τζιέσκα ως εισηγητή για τη γνωμοδότηση του Εθνομοθετήν. Ε, την βασική αρμοδιότητα, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η νομική επιτροπή. Μία αντιπροσωπεία μας με 7 μέλη ε, πήγε στην Ισπανία και συναντήθηκε με τους υπεύθυνους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ισπανίας στις 2 και 3 ε, Δεκεμβρίου εν ώψη της ε, Ισπανικής ε, Προεδρίας. Είχαμε αρκετά ενδιαφέρουσες ε, συναντήσεις και νομίζω ότι όλοι όσοι ήταν παρόντες είναι σήμερα εδώ. Υπενθυμίζουμε ότι ε, μερωθήκαμε με τον Διέγκο Λόμπε Καρίλιο, υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίο μα εξήγησε ότι η θέση σε ισχύ τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα είναι προτεραιότητα τη ε, Ισπανική Προεδρία, απόλυτη προτεραιότητα και εντόπισε τα πιο σημαντικά προβλήματα που είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπή μας. Καταρχά, η, συνεργασία με την μόνιμη Προεδρία και τις εκπεριτροπή προεδρία του Συμβουλίου η σχέση με τον πρόεδρο του Συμβουλίου και με τον είπατε εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων. Προφανώς συζητήσαμε και την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων και ο Υφυπουργό ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει διαθεσμική συμφωνία. Είναι υπέρ αυτής της ιδέας. Ένα άλλο επίγον θέμα το οποίο συζητήσαμε είναι η ολοκλήρωση του Κοινοβουλίου μέσω των πιο συγκεκριμένα των 18 μελών του ε, στο σώμα του Κοινοβουλίου και η Προεδρία της Ισπανίας ε, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ένταξη των συναδέλφων αυτών. Και σκοπεύουν να παρουσιάσουν πολύ σύντομα ένα ψήφισμα, μια έκθεση, ούτω ώστε αυτό που προβλέπει η συνθήκη να εφαρμοστεί πολύ γρήγορα με όλα τα απαραίτητα νομικά εργαλεία. Επίσης, ε, συμφωνεί η Ισπανική Προεδρία ότι η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι προτεραιότητα. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ του ΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Επίσης, συναντηθήκαμε με την Μικτή Επιτροπή ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση με υπό την Προεδρία του κ. Μίγκελ Αριέλης και την επόμενη μέρα Εγκρίθηκαν δύο τροπολογίες του Ισπανικού Συντάγματος ε, προκειμένου να, να περάσει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Κυρίως ό,τι αφορά ε, τον έλεγχο της επικουρικότητας και την, τον, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Επίσης, οι αυτόνομες κοινότητες θα πρέπει να παρέμβουν για να ελέγξουν την επικουρικότητα και καθώς και την Europol και Eurojust. Το απόγευμα της πρώτης μέρας έγινε μια συνάντηση στο Πανεπιστήμιο ε, του Σαν Πάολο με πιο γενικές συζητήσεις, αλλά υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τους φοιτητές και από τους καθηγητές και όλοι εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκφραστεί με δημοκρατικό και ενιαίο τρόπο, ενωμένο τρόπο στη διεθνή σκηνή. Ε, συνεχεία, κατά τη διάρκεια του δείπνου ε, έγινε μια συζήτηση με μια ομάδα ε, πανεπιστημιακών η ομάδα των καθηγητών από την επωνυμία Ζαμονέ. Ε, η απόψεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Καλό θα ήταν να έχουμε και ένα γραπτό κείμενο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα γραπτό κείμενο από τη συζήτηση αυτή. Γιατί νομίζω θα πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το κείμενο. Ε, στο τέλος της δεύτερης μέρας ε, συναντηθήκαμε οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών και το βασικό θέμα ήταν η εμπλοκή των πολιτών στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ενημέρωση που πρέπει να δοθεί στους πολίτες, ούτως ώστε να ενδιαφερθούν για τα θέματα της Ευρώπης. Με αυτές τις πληροφορίες νομίζω ότι εξαντλήσαμε και το σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης. Στο σημείο 3 έχουμε την έκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων που προηγήθηκαν τη σημερινή. Έχουμε τα πρακτικά της 3 ε, και 4 Νοεμβρίου 2009, 24 Νοεμβρίου 2009, και 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου του 2009. Αν κάποιος έχει παρατηρήσεις για τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων, έχει καλώς αλλιώς, θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν. Πάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ έντονο, θεσμικές πτυχές της πρόσχωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Όπως για την πράξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μία έκθεση πρωτοβουλίας για αυτό το σημείο ε, στις 17 ε, Δεκεμβρίου εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων. Ε, σε αυτή τη δουλειά ενεπλάκει και η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 50. Εγώ και ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών ε, αυτή την πρόταση. Ο συνάδελφος Γιαρέγουη ήταν ο εισηγητής. Καλό θα ήταν να εκφράσουμε τη γνώμη μας εμείς πριν το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η Κομισιόν και η Ισπανική Προεδρία θέλουν να υπάρξει απόφαση για αυτό το σημείο μέσα στο πρώτο εξάμεινο της Ισπανικής Προεδρίας, το πρώτο εξάμεινο του 2010 δηλαδή. Θα μπορούσα να δώσω τον λόγο τώρα στον συνάδελφο τον κύριο Ρέγουι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά λοιπόν βρισκόμαστε στην φάση εκπόνησης μιας έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θεωρώ ότι είναι μια από τα πιο σημαντικές, μια από τις πιο σημαντικές εκθέσεις ως έγγραφο που πρέπει να μπορέσει να αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της Συνθήκης Λισαβόνας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στο άρθρο 6 η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει όχι την βούληση αλλά την απόφαση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσχωρήσει στην Σύμβαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας αναφέρω μια σκέψη για την προέλευση, την τις ρίζες αυτού του θέματος. Όπως γνωρίζετε από την αρχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν προβλήματα ή αμφιβολίες για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε μέχρι τη δεκαετία του 70 και το επαναλαμβάνω αυτό κάποια συνταγματικά δικαστήρια και συγκεκριμένα το συνταγματικό δικαστήριο στη Γερμανία και το Ιταλικό συνταγματικό δικαστήριο στο παρελθόν δεν δεχόντουσαν, έφτασαν στο να μην δέχονται το κοινοτικό δίκαιο όταν οι αρχές ήταν αντίθετες όσον αφορά συνταγματικές αρχές για την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νομολογία που ξεκίνησε από πλευρά του 10 του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο, δηλαδή του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αυτόν τον τρόπο ένα διτό στόχο αναλαμβάνει, επομίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός να εκπονήσει μια χάρτα ξεχωριστή, εκπόνηση ξεχωριστή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των θεμελιωδών ε, ελευθεριών και δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο, ας το πω έτσι, καταλήγει στην τελευταία επισημοποίηση ε, μέσω της συνθήκης της Νίκης και εντάσσεται στη συνθήκη τώρα ακριβώς της Λισαβόνας, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 6. Και γι' αυτό λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχουμε ήδη διαμορφώσει τη δική μας χάρτα με τις τρεις εξαιρέσεις που δυστυχώς υπήρξαν σε σχέση με αυτή την χάρτα ο Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία και Δημοκρατία της Τσεχίας, οι τρεις εξαιρέσεις, αλλά ωστόσο σε σχέση με την επίσημη, ε, ας το πω έτσι, ολοκλήρωση με τη συνθήκη της Λισαβόνας, έτσι στο δεύτερο του άρθρου 6 προβλέπεται αυτό, δηλαδή ακριβώς η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και έτσι σίγουρα κάτι το οποίο είχαμε στο άρθρο 9 στο παρελθόν του συντάγματος δηλαδή που απερίφθη όμως το 2005 Θέλω να πω σε σχέση με αυτά ότι αυτή η απόφαση να ενταχθεί στη συνθήκη η προσχώρηση της ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε αυτή τη χάρτα είναι αποτέλεσμα μιας διαβούλευσης που έγινε κατά το παρελθόν ε, σε σχέση με το δικαστήριο του Λουξεμβούργου για να θεσπιστούν ποιες θα έπρεπε να είναι οι όροι και προϋποθέσεις ε, για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη σύμβαση. Και το δικαστήριο ήδη το 1996 θέσπισε, καθόρισε τις απαιτήσει, την απέτηση δηλαδή ότι ήταν αναγκαία η μεταρρύθμιση, η συνταγματική μεταρρύθμιση των συνθήκων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ένταξη αυτή τη απόφαση στο πρωτογενέ δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα με τη χάρτα άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου ε, του προηγουμένου έτους και με την προσχώρηση στην Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση όταν θα γίνει αυτή θα έχουμε ένα πλαίσιο πλέον νομικής ασφάλειας και βεβαιότητας, πλήρως ενισχυμένης και πλήρους ασφάλειας και βεβαιότητας για την εφαρμογή και υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και όλων των αρχών σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο, όλων αυτών των αρχών όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο και Πώ θα αρθρώνει λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δηλαδή των θεσμικών οργάνων. Όλα αυτά καθορίζονται. Και τώρα θα είναι αναγκαίο πλέον να υπάρξει η άρθρωση αυτή και η ένταξη μέσω των δύο αυτών προδιαγραφών, δηλαδή της, επιστολή, της χάρτας και της ε, ε, συνέλευσης, ώστε οι δύο αρχές ε, το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου να είναι τα κυριότερα όργανα. Αυτά είναι κατά η ουσία της έκθεσης αυτής. Της έκθεσης που θα υποβάλουμε δηλαδή σε αυτή την Συνταγματική Επιτροπή καταρχήν και σε σχέση με το άρθρο 50 με την παρακολούθηση από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών διαμορφώνεται έτσι, παίρνει σάρκα και οστά, παίρνει ουσία αυτή η αρχική προέλευση, αυτή η διαδρομή. Και τώρα θέλω να επισημάνω στους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής ότι για αυτή την απόφαση υπάρχουν πολλά τεχνικά και πολιτικά θέματα, σημαντικά που πρέπει να διευκρινιστούν και να επιληθούν και στην έκθεση που, θα, ε, που ε, έχουμε υποέγκριση. Πρώτα απ' όλα το θέμα πώς θα προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη σύμβαση. Προβλε, προβλέψιμο είναι και προβλέπουμε, αυτό το οποίο εξετάζουμε είναι η πιο άμεση οδός, μια συμφωνία, δηλαδή. Αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνάψει μια τέτοια συμφωνία και όλα τα κράτη-μέλη που συναποτελούν τμήμα της ε, ε, ευρωπαϊκής αυτής ε, οικογένειας. Και ταυτόχρονα θα εξεταστούν οι πιθανές τροποποιήσεις ή στη σύμβαση ή στα πρωτόκολλά της. Και θέλω να το υπενθυμίσω αυτό, συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, ότι το 8ο πρωτόκολλο τη συνθήκη Λισαβόνα, δηλαδή εκείνο το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσχωρήσει στην σύμβαση, έχει μια σειρά ορίων και μια σειρά απαιτήσεων μια σειρά διαχωριστικών γραμμών και απαιτήσεων. Συγκεκριμένα η συνθήκη τη Λισαβόνα μας επιβάλλει η συνθήκη προσχώρησης ένταξης τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή τη σύμβαση δεν θα πρέπει να τροποποιεί, να αλλοιώνει την συγκεκριμένη κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και των πρωτοκόλων καθώς επίσης και σε σχέση με κάποιες πιθανές εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις ε, που διατυπώνονται ή έχουν διατυπωθεί από κράτη-μέλη ιδιαίτερα. Αυτό τι σημαίνει, ότι η εφαρμογή, δηλαδή η υλοποίηση της ε, ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη σύμβαση θα μας θέσει νομικά προβλήματα σημαντικά όσον αφορά την εμβέλειά τους. Μια και δεν είναι βέβαιο, δεν είναι ασφαλές ότι αυτή η εφαρμογή και η υλοποίηση θα είναι καθόλου ενιαία, με ενιαία μορφή. Μια και υπάρχουν κράτη που υπάρχουν εξαιρέσεις ε, μέσω της μη αποδοχής των πρωτοκόλων ε, της σύμβασης για κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Αν υπήρχε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δεν θα είχε ας το πούμε έτσι αποδεχθεί το πρωτόκολλο όσον αφορά δηλαδή την απόρριψη της, την καταδίκη της θανατικής ποινή, θα είχαμε μια περιορισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή αυτής της αρχής για αυτό το κράτος όχι όμως για το κοινοτικό δίκαιο αλλά μόνο για αυτό το κράτος ένα ε, παράδειγμα ως ε, υπόδειγμα για να δείξω ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη σύμβαση δεν θα επιτρέψει δυστυχώς πιστεύω εγώ μια κατ' δεν θα, θα αναβληθεί κατ' εξαίρεση χαρακτήρα χαρακτήρας όσον αφορά κάποια κράτη. Μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εκείνη η οποία θα προσχωρήσει στη σύμβαση και τα πρωτόκολλα της. Όμως αυτή η σύμβαση, η προσχώρηση θα πρέπει να καθορίζει με ποια μορφή και τρόπο θα προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποια πρωτόκολλα ε, εκ Και πρέπει εδώ να επισημάνω και να πω ότι θα ήταν πιθανό σε αυτή την περίπτωση και είναι ένα από τα θέματα που τίθενται υποσυζήτηση αν αυτή η προσχώρηση θα είναι πλήρη προσχώρηση στο σύνολο των αρχών της σύμβασης και των πρωτοκόλων τη, ή όχι. Πάντα φυσικά λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να είναι σεβαστό, μια και το καθορίζει αυτό η συνθήκη τη Λισαβόνας, να είναι σεβαστό το θέμα των εξαιρέσεων που υφίστανται για κάθε κράτο μέλο ή για κράτη-μέλη. Και αυτά ήθελα επίσης να σας επισημάνω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να επιλύει αυτό το οποίο θα έπρεπε να αποκαλέσουμε την αρχή της αυτονομίας και την αρχή αυτονομίας δικαίου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πιθανότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Πιστεύω ότι ως προς αυτό θα ήταν αναγκαίο να επιστήσουμε την προσοχή και σε κάτι άλλο ότι στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου το 10 λογικό είναι ότι δεν θα χάσει την λειτουργία του ως ανωτά του δικαστή στα της νομικής δικαστικής αρχής ε, για θέματα τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν ή να προσφύγουν κάποιοι στο 10 και πιθανόν η προσφυγή κιόλας σε αυτό το 10 στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο καθώς επίσης ε, όταν θα έχουν εξαντληθεί από κρατικής πλευράς στα κράτη-μέλη οι προσφυγές στα εθνικά δικαστήρια, ε, τότε θα υπάρχει δυνατότητα άσκησης προσφυγής στο 10, στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ώστε βλέπουμε ότι το δικαστήριο του Στρασβούργου θα πρέπει να θεωρείται ένα ανώτατο δικαστικό όργανο που θα ασκεί εξωτερικό έλεγχο για τις υποχρεώσεις ε, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο για την Ένωση. Διεθνές δίκαιο και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένα τρίτο θέμα που θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και ε, θα έπρεπε να ζητήσουμε εδώ διευκρίνηση ή λύση είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θεσμικά όργανα της Σύμβασης και στο δικαστήριο. Είναι αυτονόητο φυσικά ότι κινούμε από τη βάση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσ, προσχωρώντας τη σύμβαση και όσο έχει το, το δίκαιο, να, δικαίωμα να υποβάλει έναν κατάλογο υποψηφίων για το αξίωμα των δικαστών, όπως και σε σχέση με τα κράτη-μέλη από πλευρά τους. Με αυτόν τον τρόπο αυτό είναι κάτι το οποίο μας θέτει ε, σε ισότητα όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Αλλά στο μέτρο που υπό την ξεχωριστή νομική της ε, ιδιότητα και προσωπικότητα εντάσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη σύμβαση, θα έχει δικαίωμα να έχει και εκείνη ένα δικαστή όπως τα κράτη-μέλη. Θα έχει επίσης και το δικαίωμα να συμμετάσχει όπως ε, πιστεύουμε στις συνεδριάσεις, στις συναντήσεις ε, του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν το Συμβούλιο θα ασκεί τις αρμοδιότητες του ως ελεγκτικό όργανο όσον αφορά την ομολογία και την εφαρμογή αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του 10 του Ευρωδικαστηρίου. Και επίσης θα έχει και δικαίωμα να αποτελεί τμήμα της συνέλευση που εκλέγει αυτούς. Δηλαδή εδώ τίθεται πάλι ένα πρόβλημα το οποίο θέλω να σα αναφέρω. Αυτή η παρουσία ακριβώς των ευρωκοινοβουλευτικών εκπροσώπων που θα αποτελούσαν μέρος αυτής της συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την εκλογή δικαστών είναι μόνο για αυτή την περίπτωση ή όχι. Πιθανότατα ναι, μόνο για αυτή την περίπτωση. Μια και οι δικοί μας εκπρόσωποι δεν είναι εκπρόσωποι όπως οι άλλοι μόνιμοι εκπρόσωποι που προέρχονται από τα εθνικά δικαστήρια και συναποτελούν, συναπατίζουν ε, και το, ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης που υποσυστηματικό τρόπο συζητούνται μια ολόκληρη σειρά θεμάτων μία φορά ετήσια για παράδειγμα, ας το πούμε, ε, ε, δικαστές. Εδώ τίθεται το θέμα επίσης που δημιουργεί ένα πρόβλημα, διότι αυτή η παρουσία τροποποιεί, για παράδειγμα, την απλή εκπροσώπηση όσον αφορά τους κόλπους της ε, συνέλευσης, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Τίθεται ένα θέμα της ε, εσωτερικής λειτουργίας, της ίδιας της ε, συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μια και την ημέρα που θα εκλέγονται οι δικαστές θα μπορούσαν να παρουσιάζονται εκεί κάποια, ας το πω έτσι, μέλη, βουλευτές που θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που ακριβώς θα συμμετέχει έτσι και το Ευρωκοινοβούλιο εκεί. Εδώ ανοίγει ένα σημαντικό κεφάλαιο που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αυτών των διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων με την σύμβαση. Διότι θα πρέπει να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό ποιου όρου και προϋποθέσεις θα γίνουν όλα αυτά. Τώρα σε σχέση με αυτά γνωρίζετε εσείς ότι υπάρχει μακρά και περίπλοκη σύνθετη συζήτηση στους κόλπου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Διότι μια χώρα, η Ομοσπονδία τη Ρωσίας, για παράδειγμα, δεν έχει ακόμα υπογράψει το πρωτόκολλο υπαριθμό 14. Το υπαριθμό 14 πρωτόκολλο είναι μια προσθήκη ε, όσον αφορά το, τη σύμβαση για την διευκόλυνση του δικαστηρίου που είναι υπερβολικά φορτωμένο. Έχει πάρα πολλές ε, υποθέσεις ε, και έτσι για να γίνει πιο ευέλικτο. Πρέπει επίσης μέσα στο πλαίσιο αυτών των λειτουργιών να μπορέσει να εξεταστεί το θέμα που από δικαστικής πλευράς θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη ενεργητικότητα. Και έτσι εδώ και χρόνια εδώ η προσπάθεια της έγκρισης αυτού του πρωτοκόλου εκκρεμεί. Η, ομοσπονδία, η συνομοσπονδία, η ρωσική ομοσπονδία είναι αντίθετη. Όμως ακριβώς ε, ε συμπτωματικά αυτές τις ημέρες ε, επιλύεται διότι στις 15 Ιανουαρίου πριν από λίγες ε, μέρες η Ντούμα, η Ρωσική Βουλή ενέκρινε το πρωτόκολλο υπαριθμό 14 και εκείνο που απομένει είναι η Ανώτατη Βουλή, το δεύτερο κοινοβουλευτικό σώμα, επίσης να το εγκρίνει. Εδώ ζήτησαν οι ολοκληρώσει κάτι που αφετέρου από την άλλη πλευρά υπάρχει στη σύμβαση. Η παρουσία δηλαδή ενό Ρώσου δικαστή σε αυτή την περίπτωση. Πάντα σε όλε τι περιπτώσει που θα αφορούν τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό προβλέπεται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και την λειτουργία των πραγμάτων. Και αν με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε και θα μπορούσε να διασφαλίσει σε όλα τα θέματα που εμπλέκει, εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει Ευρωπαίος δικαστής και έτσι θα απαιτήσουμε με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του δικαστή που έχει προτείνει, θα έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις υποθέσεις. Έτσι λοιπόν περιγράφω και καθορίζω τα, ε, ε, ένα πρόβλημα το οποίο τίθεται από αυτό το ζήτημα. Το επόμενο ζήτημα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω ποιο είναι. Είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στην συμμετοχή με συγχωρείτε μια στιγμή στην δυνατότητα που ίσως επίσης θα πρέπει να εξεταστεί από πλευράς μας για να μπορεί ένα κράτος μέλος να μπορέσει να υποβάλει κάποια ένσταση ή να υπάρχει κάποια αντίρρηση έναντι άλλου. Αυτό καταρχήν θα ήταν κάτι πιστεύουμε που θα παρέβαινε την συνθήκη της Λισαβόνας και δεν θα έπρεπε να δούμε πώς και γιατί θα μπορούσε κάτι τέτοιο να τεθεί. Και θα είχαμε την, ας το πω έτσι, το μη εφικτό ε, τέτοιας κατάστασης. Μια άλλη ερώτηση, ένα άλλο θέμα είναι η παθητική νομιμοποίηση. Σε σχέση δηλαδή με τα αιτήματα των πολιτών, προς ποιον θα στρέφονται όταν θα πρόκειται για την εφαρμογή μιας ρήτρα ή διάταξης σε σχέση με την παραβίαση μιας αρχής των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου ή των πολιτικών ελευθεριών. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν πάνω από τρεις δυνατότητες και εδώ θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να είμαστε, ας το πω έτσι, πλήρης στην άσκηση των δικαιωμάτων από τη Σύμβαση. Όταν ένα κράτος εφαρμόζοντας τις αρχές του κοινοτικού δικαίου βλέπουμε ότι σε σχέση με τους πολίτες ή τα θεσμικά όργανα θεωρεί ότι υπάρχει μια τέτοια παραβίαση, τότε θα πρέπει να υποβάλλεται αυτή όσον αφορά το αντίστοιχο κράτος μέλος. Όταν θα είναι ένα θεσμικό όργανο ή ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνο το οποίο ασκεί αυτές ε, τις δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, ε, τότε σε περίπτωση παραβίασης ε, θα στρέφεται το παράπονο ή προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι όταν ε, πλανάται η αμφιβολία ε, σε σχέση με την ευθύνη του ε, ποιος είναι υπεύθυνο, τότε πρέπει να καθορίσουμε την αρχή ότι ο πολίτης μπορεί να ασκήσει προσφυγή και κατά των δύο, και κατά του κράτους μέλους και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο πρόβλημα είναι εκείνο που τίθεται αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμμετάσχει ως συμβαλόμενο μέρος στις διεργασίες και διαδικασίες που θα συνεπάγεται μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να θεσπίσουμε την αρχή εδώ ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη επίσης και ιδιαίτερα εκείνα μπορούν να εντάσσονται στην διαδικασία και διεργασία αυτή όταν υπάρχει ένα άμεσο συμφέρον σε σχέση με μια τέτοια προσφυγή ή καταγγελία ή επειδή αφοράται άμεσα ένα κράτος μέλος ή επειδή ναι, μένει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ έχει ασκηθεί μια τέτοια προσφυγή κατά, του κράτους, κατά ενός κράτους μέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχει κοινοτικό συμφέρον να τοποθετηθεί και να δράσει. Εδώ μπορεί να τίθεται ένα πρόβλημα Ποιε είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι υπό τους οποίους ένα κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση συναποτελούν μέρος αυτής της διεργασία όταν δεν αφορώνται άμεσα μέσω μιας καταγγελία ή προσφυγής θα έπρεπε πιστεύω να προσπαθήσουμε να δούμε μέσα στο πλήρε πλαίσιο άσκησης δικαιωμάτων αυτή τη συμμετοχή και όχι τη συμμετοχή του ω τρίτων μερών ως τρίτων ενδιαφερόμενων μερών διότι αυτό θα ήταν διαφορετικό εδώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να υπάρξουν, πώς να το πω μια στιγμή, διαφορές που θα απορρέουν μεταξύ του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και του 10 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Λοιπόν, εδώ εγώ πιστεύω ότι αυτή η ε, διαδικασία πρέπει να καθιστά σαφές ότι πρέπει να εξαντλούνται πρώτα όλα τα δικαστικά μέσα για να καταλήγει κάποιος στο Στρασβούργο. Και όταν καταλήγουμε σε κάποιες ε, νομοθετικές, νομολογικές ρυθμίσεις που μπορεί να θεωρηθούν αντιφατικές ή να δημιουργούνται τριβές, το σημαντικό είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των δύο δικαστηρίων για την εξέβρεση μιας λύσης Παρότι εγώ πιστεύω προσωπικά ότι η σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση αυτή καθορίζει, προσανατολίζει την ερμηνεία αυτής της χάρτας και εδώ στο πλαίσιο η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών μπορεί να τοποθετηθεί πιο εξειδικευμένα για αυτές τις πιο στενές ε, περιπτώσεις ή έννοιες ε, ε, αυτών των θεμάτων. Όμως, σε σχέση με την συνέλευση ε, που ε, έχει αρμοδιότητα ερμηνείας αποτελεί πηγή η σύμβαση αυτή για την ε, ερμηνεία και την εφαρμογή της, των αρχών της σύμβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο πριν αναφέρθηκα στο πρωτόκολλο υπαριθμό 14. Εμείς πρέπει να επιστήσουμε επίσης την προσοχή εδώ ότι η διαπραγμάτευση για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει σε σχέση με ένα λειτουργούν δικαστήριο που θα λειτουργεί θετικά και έτσι, αν επιληθεί το θέμα της προσυπογραφής, της επικύρωσης του πρωτοκόλου υπαριθμών 14 τις επόμενες ε, ημέρες ή εβδομάδες, θα έχουμε ένα δικαστήριο μπροστά μας που θα έχει επιλύσει ένα από τα μείζωνα θέματα που αντιμετωπίζει. Αυτό το πρωτόκολλο 14 είναι συνέχεια άλλου που υπήρξε κατά την δεκαετία του 90, αλλά που δεν δημιούργησε τις επιθυμητές ε, επιπτώσεις ε, και όρους και προϋποθέσεις. Και έτσι λοιπόν είδαμε ότι όλα αυτά δεν μπόρεσαν να επιλύσουν το, τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, τεράστιο φόρτο εργασίας που έχει το δικαστήριο, που έχει μια πολύ σημαντική δομή, όμως λαμβάνοντας υπόψη την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη σύμβαση, με όλες τις δυνατότητες ε, διάνοιξης, δυνατότητας άσκησης προσφυγής ε, από πολίτες, ε, πρέπει οπωσδήποτε να επιληθεί αυτό το θέμα, να έχει επιληθεί προηγούμενα πριν από την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και μια τελευταία ε, παρατήρηση, μια τελευταία σκέψη, πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η απόφαση ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην σύμβαση αυτή. Τέσσερις προϋποθέσεις είναι αναγκαίες πιστεύω εγώ. Πρώτον η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεύτερον, μια απόφαση ομόφωνη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τρίτον, μια διαπραγμάτευση για μια συμφωνία προσχώρησης με την Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τέλος, τέταρτο, έγκριση από τα κράτη-μέλη όσον αφορά το συνταγματικό πλαίσιο από πλευρά τους. Με αυτούς τους όρους και με αυτούς τους άξονες θεωρώ ότι έχω περιγράψει τα μεγαλύτερα θέματα τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει αυτό το χαρτοφυλάκιο, αυτό το ζήτημα. Θέλω να σας επισημάνω ότι με την ε, ένδειξη του Προέδρου η πρώτη συζήτηση σε σχέση με αυτό ε, θα είναι ο επόμενος μήνας ε, του Φεβρουαρίου και θα έχουμε, έχουμε και υπόψη τη διεξαγωγή μιας ακρόασης για να υπάρξει μια συνάντηση σαν αυτή που είχε συμφωνηθεί στην σύνοδο συνάντηση των συντονιστών. Δηλαδή να καλέσουμε πέντε ή έξι ε, εμπειρογνώμονες ε, για παράδειγμα από το δικαστήριο ή από το δικαστήριο συνταγματικό, ε, με συγχωρείτε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Στρασβούργου ή από το ΔΕΚ για να κάνουμε μια ακρόαση από κοινού μαζί τους, να ακούσουμε τις απόψεις τους και να θέσουμε τις ερωτήσεις μας. Και έτσι στη συνέχεια το Μάρτιο, Απρίλιο μπορούμε να δούμε, να τροποποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την έκθεση. Αυτά είναι όλα όσα είχα να σας πω. Είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις παρατηρήσεις σας για να βελτιωθεί ακόμα περαιτέρω αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γιαουρέγουι Ατόντο. Πολλά είναι τα προσεπίληση θέματα, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε πολύ σοβαρά, ακριβώς για να τα επιλύσουμε. Και αν συμφωνούν και οι συντονιστές, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και μια ακρόαση, όπως είπατε κι εσείς. Ο κ. Σεβερίν είναι ο πρώτος συνάδελφος που θα μιλήσει, αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να σας προκαλέσω εγώ. Πρώτον, η σχέση μεταξύ ΔΕΚ και Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Το δικαστήριο του Στρασβούργου ε, προβλέπει ότι δεν μπορούν να γίνουν παραδεκτές υποθέσεις αν δεν έχουν εξαντληθεί, δεν έχουμε εξαντληθεί εσωτερικές οδοί. Όπω είπε και ο κ. Ιγιαρέουι, το, το δικαστήριο του Στρασβούργου είναι ένα επιπλέον βήμα μετά τις διαδικασίες των κρατών. Αν όμως τα θέματα αφορούν τα ανθρώπινα, αν λοιπόν τα θέματα αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει πρώτα να έχουμε εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα στα κράτη-μέλη και μετά να φτάσουμε στο Στασβούργο. Αυτό είναι το απότατο βήμα. Έτσι. Μια άλλη παρατήρηση, έτσι λίγο προκλητική αν θέλετε, για τις εξουσίες του Κοινοβουλίου κτλ. Το παράδοξο είναι, είναι ότι όπως έχουν σήματα τα πράγματα ε, με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση προβλέπεται ότι θα επικυρωθεί και θα εφαρμοστεί για όλες τις χώρες που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει μόνο στη Σύμβαση όχι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί αν ήταν έτσι, θα έπρεπε απλώς να τροποποιήσουμε το αρμόδιο άρθρο που προβλέπει τα της ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Εμείς δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Ε, τώρα, όλες οι πράξεις που αφορούν τη λειτουργία του δικαστηρίου είναι κάτι το τελείω διαφορετικό. Έτσι. Αλλά αυτό το είχε πει και ο συνάδελφος ε, Γιαρέγουι, ο κ. Σεβερίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από λίγα χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση, εγώ ανήκα στην ομάδα των συναδέλφων που ήταν πολύ υπέρ της ιδέας της ένταξης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτήσει την νομική προσωπικότητα. Ε, Ακούγοντα τώρα τα σχόλια του Ισπανού συναδέλφου, διερωτώ με αν πράξαμε καλώ. Γιατί αυτή η δουλειά ε, προποθέτει πολλή προσπάθεια. Ή μήπω δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Ε, γιατί τελικά δημιουργούμε πάρα πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα που ήθελα να θίξω, εν μέρη τα θίξατε εσείς κύριε Πρόεδρε. Α ξεκινήσω όμω με το τελευταίο τμήμα τη έκθεσης, με το τέλο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συναντηθούμε με του εμπειρογνώμονε, να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση, δηλαδή υποστηρίζω αυτή την πρόταση του κυρίου Γιουρέγουη. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό θέμα το εξή. Δεν υπάρχει πραγματική πρόσβαση στη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, αν δεν δεχτούμε και τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Και αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο βήμα προσφυγής αυτή τη στιγμή όλα τα, μόνο όταν όλα τα εθνικά ε, βήματα δικαιοδοσίας έχουν εξαντληθεί και όλα τα ε, ε, εθνικά ενδικά μέσα έχουν εξαντληθεί. Επομένως, όχι το Στρασβούργο του Λουξεμβούργου, αλλά το, Στρασβούργο, το δικαστήριο του Στρασβούργου θα έχει τον τελευταίο λόγο. Έτσι, αν κατάλαβα καλά. Το σημείο 3 τώρα που θέλω να αφήξω. Θα γίνουμε συμβαλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως ε, απόρρια του γεγονότος ότι έχουμε αποκτήσει τώρα νομική προσωπικότητα. Επομένως, θα μπορούμε και να μηνύουμε στο δικαστήριο, να μας μηνύουν στο δικαστήριο, μόνο σε ό,τι αφορά τις πράξεις και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των κρατών μελών της. Τέταρτο σημείο. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επικυρώσουν την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Γιατί τα κράτη-μέλη επικύρωσαν τη συνθήκη της Λισαβόνας ήδη. Επομένως συμφώνησαν ότι θα γίνουμε και συμβαλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και ε, κάτι άλλο αυτός που θα γίνει μέλος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομική οντότητα. Αντίθετα τώρα, οι χώρες, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα κράτη θα πρέπει να επικυρώσουν την προσχώρηση αυτή. Γιατί, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, Οι κανονισμοί του, Ευρωπαϊκού, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συγγνώμη λένε, ότι πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Επομένως, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να κάνουν αυτή την, α, την επικύρωση. Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μας μηνύσουν γιατί παραβιάζουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και πρέπει να σκεφτούμε αν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά μας δικαστήρια, αν χρειαστεί. Τώρα, θα ήθελα να τελειώσουμε την εξή παρατήρηση. Ξέρω ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο εισηγητής μας θα πρέπει να σκεφτεί το θέμα της ενότητας της δικαιοδοσίας ε, στην Ευρώπη και την ενότητα των κανονισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί αν λόγω, για λόγους ουσίας ή λόγω νομολογίας υπάρχει ε, σύγκρουση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ε, και της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τότε μπορούμε να έχουμε σοβαρότατα προβλήματα και μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις à la carte στους ενδιαφερόμενους. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι αποδεκτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τα θέματα των συμβάσεων, όχι της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, των υπολείπων. Για να δούμε πώς μπορούμε να ενοποιήσουμε τη δικαιοδοσία, αν υπάρχει σύγκρουση δικαιοδοσίας, πώς μπορούμε να ενοποιήσουμε το ουσιαστικό δίκαιο και να προσπαθήσουμε να επινοήσουμε κάτι ώστε να διευκολύνουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μια και το δικαστήριο αυτό κινείται πάρα πολύ αργά, δουλεύει πάρα πολύ αργά γιατί κατακλείζεται από υποθέσεις και αν προσφύγει και ένα, ενταχθεί και ένα νέο μέλος ε, τη λόγω σύμβασης ε, θα κατακλειστεί ακόμη περισσότερο από υποθέσεις από ό,τι σήμερα. Να υπογραμμίσουμε πόσο περίπλοκο αλλά και πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό το θέμα από νομικής πλευράς. Ε, θα το υπογραμμίσει ακόμη περισσότερο ο κύριος Μέντες Δεβίγκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ Χαίρομαι ιδιαίτερα που γίνεται αυτή η συζήτηση, καθώς και για την απόφαση της Επιτροπής μας να λάβει την πρωτοβουλία και να εκπονήσει την έκθεση αυτή. Συγχαίρω τον εισηγητή. Και θα ήθελα εξ αρχής να κάνω μία δήλωση αρχής. Δεδομένου ότι είμαστε στο ίντερνετ θα ήθελα σαφώς να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δεν είναι επειδή τώρα θα αρχίσουμε να τα σεβόμαστε επειδή θα συνυπογράψουμε αυτή τη σύμβαση, το κάνουμε ανέκαθεν. Είναι αλήθεια ότι δεν προβλεπόταν ο χάρτης, αλλά μετά από την μέρα όπου υπογράφηκε και προβλέφθηκε η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στη δεκαετία του 60 και του 70, μεριμνήσαμε για τη δέσμευση της στήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Σύμβαση της Ρώμης, η Σύμβαση του 50, Το 1987 ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος ε, Ορέχα και ο πρόεδρος του Συμβουλίου ήδη είχε υπογράψει μια συμφωνία σε σχέση με την ε, υπογραφή της σύμβασης αυτής. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Μετά έγινε η έκθεση του κυρίου Ντεγκούχτ και στη συνέχεια το Μάστριχτ μετά στη συνέχεια το άρθρο 16.2 που αναφερόταν σε αυτό, αλλά θεωρήσαμε πως όλα αυτά δεν αρκούσαν και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την πρωτοβουλία και ε, συγκάλεσε αυτή τη συνέλευση που συνέταξε τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι δραγμένος στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και εδώ θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πιστεύω πως ε, καταρχήν, όχι πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη σύμβαση της Ρώμης και τον χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Οι μεταβατικές και οι οριστικές διατάξεις ε, ορίζουν ότι κάθε αναγνωρισμένο δικαίωμα στον χάρτη θα ε, εφαρμόζεται σύμφωνα με στην Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση με επιφυλάξει των κρατών μελών σε σχέση με συγκεκριμένα δικαιώματα. Και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στον χάρτη των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελεί τμήμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Άρα η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Ο κύριος Σεβρέα έφυγε, όχι, είναι εδώ στην αίθουσα έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα. Ενεργήσαμε σωστά ή όχι. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει αμφιβολία πως σωστά ενεργήσαμε. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση αποτελεί ένα βήμα προόδου σε σχέση με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αυτό το ζητούν οι πολίτες και αποτελεί μια επιπλέον εγγύηση. Άρα λοιπόν σωστά ενεργήσαμε. Τώρα θέλουμε να λύσουμε τα νομικά ζητήματα. Είναι ένα καθόδε ζήτημα και δεν θα πρέπει εδώ να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η διακυβερνητική διάσκεψη και ίσως εδώ να Έχασα εγώ κάπως ε, τον ε, λογαριασμό σε σχέση με αυτήν τη διακυβερνητική διάσκεψη. Πάντως μετά από την συνταγματική συνθήκη φτάνουμε στο εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει με ειδική πλειοψηφία, ΣΑΛ, μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών των στοιχείων που οδήγησαν στο ότι χρειάστηκε να τροποποιήσουμε την ειδική πλειοψηφία, να αντικαταστήσουμε μάλλον την ομοφωνία από την ειδική πλειοψηφία. Ε, ε, έχουμε αυτό το ρήμα το «σαλ» που σημαίνει «οφείλει» και όχι «με ή δύναται». Ε, και πιστεύω πως από εδώ και μπρος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που στην πλειοψηφία του θεωρεί πως είναι θεωρεί αυτή η εξέλιξη, θα μπορέσει όντως να προχωρήσει, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια σημεία προς ρύθμιση και τα κράτη που δεν επιθυμούν να το κάνουν αυτό μην το αμφιβάλλετε, θα ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση για να δείξουν ποιες είναι οι δυσκολίες νομικής φύσης που όντως υπάρχουν. Νομίζω πως η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου θεωρεί πως είναι καλή η επιλογή. Η ομάδα μου το πιστεύει επίσης και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιληθούν όλα αυτά τα ζητήματα που είναι δύσκολα στην επίλυσή τους και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια τροχοπέδη αυτό είναι ο στόχος αυτή τη έκθεσης. Εγώ συμφωνώ για την διεξαγωγή μιας ακρόασης. Θα μπορούσαμε ίσως να καλέσουμε έναν άνθρωπο που στο παρελθόν μας βοήθησε πολύ και που ήταν και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνόδου. Είναι ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση του ζητήματος. Έχουμε τον Ρενέ Βαντερλίνγκ, σίγουρα θα τον γνωρίζετε και μαζί του είχαμε πολλές συζητήσεις για τις πρακτικές εφαρμογές, όπως είπε και ο κύριος Χαουρίκη, ε, τις πρακτικές εφαρμογές της ε, προσχώρησης στη σύμβαση. Το είπατε και προηγουμένως ότι αυτή η σύμβαση δεν αναφέρεται παρά στα κράτη-μέλη. Δεν προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια διεθνής οργάνωση θα είναι μέλος. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν τροποποίησεις και στην ίδια τη σύμβαση. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με μια διμερή απόφαση. Από τη μια πλευρά έχουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης με την σύμβασή του και από την άλλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε μόνο εμείς δηλαδή που θα αποφασίσουμε ε, θα πρέπει να γίνει η τροποποίηση και της σύμβαση. Αυτό, περί αυτού δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία και ε, ως εκ τούτου θα πρέπει να την εγκρίνουν αυτή την τροποποίηση και τα 47 μέλη του Συμβουλίου. Δεν γνωρίζω όλες τις νομικές λεπτομέρειες, αλλά η δική μου διέστηση μου λέει πως η επικύρωση θα πρέπει να γίνει από πλευράς όλων των συμβαλωμένων μερών. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα θέματα που ανέφερε ο εισηγητής μας είναι σημαντικά, αλλά το πιο ενδιαφέρον κατά τη δική μου άποψη είναι η δυνατότητα να κάνουμε μία, μία τελευταία προσφυγή στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί ε, μία προστιθέμενη αξία για τον πολίτη ή για μια ομάδα πολιτών ε, και είναι μία προστιθέμενη αξία της ε, σύμβασης. Είναι μάλιστα ένα τμήμα της αποτυχίας. Δηλαδή οι Ρώσοι πολίτες κάνουν προσφυγές καθημερινά. Αυτό οφείλεται στο ρωσικό σύστημα. Υπήρχε και ένα ήταν μάλλον και βρετανικό το πρόβλημα. Ε, παλαιότερα οι πολίτες είχαν ε, πρόσβαση στο δικαστήριο του Στασβούργου και άρα αυξανόταν πολύ ο φόρτος εργασίας του δικαστηρίου. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να ρυθμιστεί και η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να βοηθήσει στη ρύθμιση αυτού του προβλήματος. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την προσχώρηση δηλαδή για να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα. Έχω την εντύπωση κύριε Πρόεδρε πως αυτή η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση ως ε, τελευταία μάλλον ε, δυνατότητα πρόσβαση στο δικαστήριο είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα στοιχείο κλειδί αυτό. είναι ένα δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό υιοθετήθηκε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όταν γίνεται λόγος για εθνικά δικαιώματα, ακόμα και αν η προέλευσή τους είναι κοινοτική φύσης, αυτά ε, είναι στη δικαιοδοσία του εθνικού δικαίου και ήδη μπορεί κανείς να προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Πρόκειται δηλαδή για αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Νομίζω λοιπόν πως αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το προσέξουμε και να το εξετάσουμε. Δηλαδή ποιος αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχουμε κάποιο δικαστή. Ε, ε, ε, είναι πολύ περίπλοκα αυτά τα ζητήματα κύριε Πρόεδρε. Ωστόσο, θα ήθελα να επαναλάβω την άποψη της πολιτικής μου ομάδας, ότι δηλαδή είναι ένα θέμα πολιτικής σημασίας, ύψης της πολιτικής σημασίας. Από τη συνθήκη του Σπινέλη, μέχρι σήμερα και η συνθήκη του Σπινέλη το προέβλεπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν ε, θεωρούσε αυτό το θέμα ιδιαίτερα προσφυλές και ακόμα και αν είναι δύσκολο και περίπλοκο εγώ χαίρομαι που έχουμε να το αντιμετωπίσουμε και πάλι και επίσης επειδή δική μας Επιτροπή είναι αρμόδια και με εντυπωσίασε που η Νομική Επιτροπή δεν εκτίμασε κάποια έκθεση από αυτό δεν ξέρω αν είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που ανέλαβε τις αρμοδιότητες της Νομικής Επιτροπής αλλά κύριε Πρόεδρε ίσως και η Νομική Επιτροπή να πρέπει να εκφραστεί για το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω πως ε, η Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία για να ανοίξει το δρόμο για την εξέβρεση μιας τέτοια μιας λύσης. Είναι μια πρωτοβουλία εξαιρετικά σημαντική και κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα το συζητήσουμε και θα εργαστούμε σκληρά ώστε να βρούμε καλές λύσεις. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όταν μπήκα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν πολλά χρόνια, ε, η, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων λεγόταν Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για τα Δικαιώματα των Πολιτών. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ. Ehm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτές τις σκέψεις για τη σημασία του θέματος. Συμφωνώ επίσης ότι τίθενται και μια σειρά νομικά ζητήματα και προβλήματα. Πριν μιλήσουμε για αυτά όμως θα ήθελα να πω δύο λόγια για ένα κρατός μέλος και που θέλει να έχει το δικό του δικαστή σε αυτό το τομέα. Αν επαναδιοριστεί ο δικαστής αυτός, η κυβέρνηση που διορίζει αυτό τον δικαστή θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, πώς εκφράστηκε ο δικαστής αυτός για τη χώρα του, για τη χώρα μου συγκεκριμένα, τη Δανία. Η χώρα μου ε, σύρθηκε στο δικαστήριο, υπάρχει ένας δικαστής ο οποίος μιλάει για τη Δανία και η δανέζικη κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει για, τα επόμενα, για την καριέρα αυτού του ανθρώπου για τα επόμενα 7 χρόνια. Νομίζω, ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να μπλέκουμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα πρέπει μια χώρα να μπλέκεται στην, ε, στην καριέρα ενός δικαστή από την ίδια χώρα. Έπειτα, κάποια άλλα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Στη συνθήκη προβλέπεται ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της χάρτας ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και της σύμβασης. Νομίζω στο σημείο 72 λέμε ότι η χάρτα θα πρέπει να επιτρέπει να υπερασπιστούμε καλύτερα τα δικαιώματα από τη σύμβαση. Αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, γιατί η χάρτα είναι υπερεθνική, ενώ η σύμβαση είναι μια συμφωνία μεταξύ κρατών. Αν παραβιάσουμε τη χάρτα, αν επιβάλλονται πρόστιμα, τότε θα πρέπει να σεβαστούμε τη χάρτα. Ενώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης τα πράγματα συμβαίνουν διαφορετικά. Ε, νομίζω ότι έχουμε καλύτερη προστασία αν περάσουμε από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου παρά από το δικαστήριο του Στρασβούργου. Ε, υπάρχουν προβλήματα και για τις προσφυγές. Υπάρχουν επίσης και κάποιες τυπικές δυσκολίες. Το γεγονός ότι έχουμε αποφάσεις ε, δεσμευτικές από τη μία πλευρά αλλά μη δεσμευτικές από την άλλη. Το γεγονός ότι στο ΔΕΚ θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της ε, επικουρικότητας ενώ στο Στρασβούργο έχουμε μια δυνατότητα, μια ευχαίρεια εκτίμησης ε, μας δίνει μια τελείως διαφορετική ελευθερία για να οριοθετήσουμε τα νομικά θέματα. στο Στρασβούργο ε, το, Στρασβούργο, το δικαστήριο του Στρασβούργου μπορεί να εκτιμήσει ότι κάποια θέματα εκφεύγουν τη αρμοδιότητά του, που με βάση το 10 ε, είναι θέμα επικουρικότητα. Και το σημείο 72 δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην ανάπτυξη τη χάρτα. Πώ θα επιλύσουμε ένα πρόβλημα αν η σύμβαση του Στρασβούργου ε, πριτανεύει σε σχέση το δικαστήριο του Στρασβούργου προετανεύει σε σχέση με το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Μπορεί ένα πολίτη να κάνει μια προσφυγή περνώντα μέσα από τα εθνικά δικαστήρια, εν συνεχεία πάει στο ΔΕΚ που τον δικαιώνει και για λόγους καθαρά τυπικούς το καταδικασμένο κράτος να στραφεί στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έχει όμως ε, την απόλυτη ισχύ ε, και πρωτοκαθεδρία και θα του δώσει δίκιο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αποφάσεις τις δεσμευτικές και μη δεσμευτικές και θα πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα, τη δυνατότητα ε, εκτίμηση και την ευχαίρεια εκτίμηση στο δικαστήριο του Στρασβούργου σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής επικουρικότητας στο 10. Εγώ φαντάστηκα ότι τέτοιου τύπου προβλήματα θα προκύψουν όταν ε, συζητήσουμε για αυτό το πρόβλημα. Και όπως είπε και ο κύριος ε, Μέντες Τεβίγκο, Υπάρχει και το θέμα της εκπροσώπησης των κοινωνικών θεσμικών οργάνων στα πλαίσια της σύμβασης. Προσοχή, προσοχή. Ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουμε κάποιους ε, συναδέλφους από την Ανατολική Ευρώπη που με κάθε ευκαιρία όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε τη σύμβαση ε, προσπαθούν να παρακολύσουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό διαπιστώσαμε στα πλαίσια του πρωτοκόλλου 14. Συνέβη κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να διωτηθούμε μήπως χρειάζεται ένα πρωτόκολλο 15 ή μια πλήρης τροποποίηση της σύμβασης αυτή του, του Στρασβούργου. Γιατί όπως κάναμε για τη Δούμα ε, πρωτόκολλο 14 υπάρχουν τόσα τεχνικά προβλήματα που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την, α, ε, τις εργασίες μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας προειδοποιήσω όπως είπε και ο κύριος Μέντες Τεβίγκο, ε, το να τροποποιούμε μονομέρως τα πράγματα είναι επικίνδυνο. Όχι γιατί δεν έχει τη βούληση η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη, που είναι πολύ σημαντικά εξάλλου, που θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που έχουν σε πολιτικό επίπεδο. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Δεν πρέπει να έχουμε διαφορετικές νομικές διατάξεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα πρέπει ως πολίτες να θέσουμε ή ως κράτη ε, να θέσουμε το ερώτημα πού πρέπει να προσφύγουμε. Θα πρέπει αυτό το σύστημα να συγκλίνει και να μην αποκλίνει. Αυτό το σύστημα που πάμε να δημιουργήσουμε. Ευχαριστώ. Um, Uh, Πρόεδρε, συμφωνούμε όλοι πως είναι εξαιρετικά σημαντικό και συναρπαστικό ζήτημα. Αλλά θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε πως ήταν ε, ένα δούνε και λαβίνε ότι ο χάρτης αυτής θα ήταν ε, δεσμευτικός. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σταθερό για αυτό το θέμα παρά το σύμπλεγμα των περίπλοκων ζητημάτων που παρουσιάζονται στην αρχή αυτής της ε, διαδικασίας. Ο χάρτης είναι ο τρόπος να εκφράσουμε να διατυπώσουμε το, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, είναι ευρύτερο το πεδίο εφαρμογής. Όμως, οι περιορισμοί για το πώς εφαρμόζεται ο χάρτης στα κράτη μας εφαρμόζονται, ισχύουν μάλλον, και για τον χάρτη καθώς απορρέει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι αλήθεια ότι θα υπάρξουν κάποιες αντιφάσεις, ίσως και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, καθώς εφαρμόζεται για κάποιο εσωτερικό ζήτημα εντός δηλαδή των κρατών μελών και της εφαρμογής του από τις Βρυξέλλες, για να το πω έτσι. Αλλά η ένταση αυτή δεν μπορεί παρά, είναι, να είναι δημιουργική. Και για όσους φοβούνται ότι θα υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στα δικαστήρια, νομίζω πως υπερβάλλουν. Στο παρελθόν υπήρξε εντατική συνεργασία ανάμεσα στα δικαστήρια και θα πρέπει να θεωρήσουμε το Στρασβούργο ως έναν εξωτερικό επόπτη του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου και όχι ως ένα αριοπάγο. Δεν νομίζω πως αυτό θα ήταν το σωστό, η σωστή περιγραφή για το Στρασβούργο. Και επειδή το Στρασβούργο έχει τις ρίζες του στον τομέα του θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ορισμένα από τα προβλήματα που προβλέπονται αυτή τη στιγμή δεν νομίζω πως καν θα προκύψουν στην πράξη. Αν όντως καταφέρουμε να έχουμε την ε, πρόσβαση θα είναι για μας μια όθηση για τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου του Στρασβούργου γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή επιβαρύνεται από διαδικασίες και σορευμένες υποθέσεις που, με τις οποίες παλεύει να διεκπαιρεώσει. Εμείς λοιπόν μπορούμε να προσφέρουμε στο δικαστήριο του Στρασβούργου μια όθηση, ένα κίνητρο για μεταρρύθμιση και πιστεύω πως και αυτό θα πρέπει να τονιστεί στην απόφαση του Κοινοβουλίου για το θέμα. Σας ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο ο συνάδελφος Μπρόντς. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι γενικό κανόνα στην πολιτική πω δεν υποβάλλει ερωτήσει εκτό και αν ήδη ξέρει την απάντηση. Ωστόσο, εγώ θα υποβάλω ερωτήσει για τι οποίε δεν έχω την απάντηση. Η σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ το Συμβούλιο τη Ευρώπη και τη σύμβασή του θα είναι παρόμοια με αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από το 2000, δηλαδή θα έχουμε υπογράψει επί των αρχών χωρίς όμως να αποτελέσει η σύμβαση κομμάτι τη Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ή αυτομάτως θα γίνει τμήμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ε, ο χάρτης θέλω να πω, ναι. Όλες οι μελλοντικέ νομοθεσίες της Ένωσης θα ε, συνοδεύονται από κάποιο είδος εγγράφου της Κομισιόν που λέει ότι αυτή η νομοθεσία είναι συνεπής ή θεωρείται πως είναι σύμμορφη προς τη σύμβαση. Τρίτον, ένας διεθνής οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπει σε έναν διεθνό, άλλο διεθνή οργανισμό, δηλαδή το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θεωρούμε πως αυτή η δεύτερη, οι αρχές αυτού στη σύμβαση θα έχουν υπεροχή υπέρ του, δικής, του δικού μας χάρτη. Τέταρτη ερώτηση και εδώ έχω μια όριστη μνήμη ότι κάτι έχω ακούσει ίσως σε κάποια άλλη αφορμή σε αυτή την Επιτροπή στη ΛΥΜΠΕ ότι είναι δυνατόν οι τρεις χώρες που έχουν το opt-out από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί στο μέλλον να είναι σε θέση να φέρουν μια υπόθεση στο Συμβούλιο Τη Ευρώπης στο Στρασβούργο, ώστε να αμφισβητήσουν αυτά τα opt-out. Κάποιος είχε πει τη γνώμη του από αυτού, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και μια τελευταία ερώτηση που θέλω να υποβάλω. Κατάλαβα σωστά ότι δύο χώρες και οι δύο από αυτές ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπορούν η μία να προσφύγουν έναντι της άλλης στο Στρασβούργο, αλλά τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα να πάνε στο δικαστήριο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να τα πάνε τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Αυτό κατάλαβα να λέτε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μορέιρα. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο από αυτή την πρώτη συζήτηση για την πιθανή προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, συγχαρητήρια κύριε Γιαουρέγκουι για τη θαυμάσια εισαγωγή στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε Είμαι καθηγητής συνταγματικού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πανεπιστήμιό μου και επί δεκαετίες τώρα ήμουν υπέρ της ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με μεγάλη χαρά λοιπόν συμμετέχω σε αυτή την πρώτη συζήτηση. Κατά την άποψή μου η προσχώρηση, η πιθανή προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χάρτα του Στρασβούργου σημαίνει δύο πράγματα. Καταρχάς, η χάρτα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης θα γίνει τμήμα του νομικού δικαίου, του νομικού ορίζοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχει πρωτοκαθεδρία ε, έναν του δικού μας δικαίου. Γιατί για τα ανθρώπινα δικαιώματα η σύμβαση έχει ισχύ και θα είναι το υπέρτατο δίκαιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να το σέβονται αυτό. Δεύτερον, κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει τη δυνατότητα να κάνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου εναντίον οποιασδήποτε απόφαση, είτε του νομοθετικού οργάνου είτε των ε, διοικητικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δικαστηρίου, του ΔΕΚ δηλαδή, που κατά την άποψή του συνιστούν παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όλα τα θεσμικά όργανα και το δικαστήριο θα πρέπει να σέβονται την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Βέβαια δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταρχήν. Το ίδιο ισχύει στη σχέση των δικών μας συνταγμάτων και της Ευρωπαϊκής ε, Σύμβασης και δεν μας εμποδίζει, δεν εμποδίζει οι χώρες μας ε, να καταδικαστούν πολλές φορές, ορισμένες περισσότερες από άλλες, για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Επομένως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να δεχτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταδικαστεί από το δικαστήριο του Στρασβούργου είτε μέσω κανονισμών ή μέσω διοικητικών αποφάσεων ή μέσω αποφάσεων του ίδιου του δικαστηρίου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, την οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε, δεν μπορούμε να εξαλείψουμε. Επομένως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα πρέπει να προβλέψουμε να, την εφαρμογή των μέτρων που θα αποφασιστούν εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από την αρχή. Πώ θα προετοιμάσουμε τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή και την εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Γιατί ε, σε περίπτωση που υπάρχει καταδικαστική απόφαση για να εφαρμοστεί αυτή, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσουμε απλώ κάποια πρόστιμα ή κάποια οικονομική αποζημίωση. Μπορεί να σημαίνει αυτό την αναθεώρηση κάποιων νομοθετημάτων ή την αναθεώρηση των αποφάσεων του ίδιου του δικαστηρίου, ε, δηλαδή του ΔΕΚ. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι για να εφαρμόσουμε και να εκτελέσουμε οποιαδήποτε καταδίκη ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γεουρέγουη για την ενδιαφέρουσα εισαγωγή του. Εγώ δεν έχω αποφασίσει για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρώντα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα θετικό βήμα ή όχι. Υπάρχουν πρακτικά ερωτήματα τα οποία θα ήθελα για να μπορέσω να αποφασίσω να μου απαντηθούν. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξή. Με ποιον τρόπο η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βελτιωθεί. Δηλαδή, θα αλλάξει κάτι. Μήπως απλώς ε, προσθέτουμε στρώματα νομικής ε, περιπλοκότητας που θα χαροποίησει τους νομομαθείς, αλλά κανέναν άλλον. Ή θα υπάρξει πραγματική βελτίωση για το λαό της Ευρώπης, ε, για τους πολίτες της Ευρώπης. Αυτό δεν το ξέρω και θα ήθελα να μου το απαντήσει κάποιος. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα, επηρεάσει, θα επηρεαστεί μάλλον η εφαρμογή των αποφάσεών της. Δηλαδή ποιος εφαρμόζει την απόφαση εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παραβιάζει κάποιες διατάξεις. Και θα αλλάξει ο τρόπος εφαρμογής εάν κάποιο κράτος μέλος ε, θεωρείται ότι έχει παραβιάσει κάποια διάταξη. Υπάρχει απώλεια κυριαρχίας ή όχι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια κρόση και νομίζω ότι και ελπίζω να ακουστούν διάφορες απόψεις σε αυτή την ακρόση. Αυτό που δεν θέλουμε είναι μια διαδοχή ομιλητών οι οποίοι ξέρουν πολλά πράγματα και λένε όμως το ίδιο πράγμα. Θα λένε, δεν θέλω να ακούω όλους να λένε ότι πρέπει να ενταχθείτε και καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ακούσω και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Γιατί αλλιώ δεν έχει νόημα να γίνει αυτή η ακρόαση. Επομένω, αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ και περιμένω με ενδιαφέρον να δω πώ θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Χοφμάιστερ, ζητάει το λόγο. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για την Επιτροπή θα θέλαμε να εκφράσουμε βαθιές ευχαριστίες στον εισηγητή κύριο Χάουρεγγι γιατί με τέτοιο εξαιρετικό τρόπο παρουσίασε σήμερα τεχνικά θέματα τα οποία <clears throat> αφορούν αυτό το χαρτοφυλάκιο, αυτό το θέμα. Θα ήθελα σύντομα κάποιες διαργασίες να σκιαγραφήσω διαδικαστικά θέματα ή διαβήματα όσον αφορά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ήδη εσείς είπατε κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος Μπαρόζο ήδη δημόσια έχει δηλώσει ότι προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση θα είναι προτεραιότητα της δεύτερης θητείας της Επιτροπής Μπαρόζο και γι' αυτό αναμένουμε μια επίσημη τυπική σύσταση θα υποβληθεί στο Συμβούλιο όσον αφορά την έγκριση αυτών των διεργασιών αμέσως μετά την έγκριση της Επιτροπής Μπαρόζο είναι λοιπόν διατεθειμένη να υποβάλει <clears throat> μετά τις 9 Φεβρουαρίου μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ευελπιστούμε. Δεύτερον, όσον αφορά τις διαβουλεύσεις όπως όλοι γνωρίζετε υπό την συνθήκη της Λισαβόνας θα ενημερώνεται πλήρως και θα εμπλέκεται το Ευρωκοινοβουλίο και προσβλέπουμε στο να υλοποιηθεί το σχετικό άρθρο <clears throat> για την εμπλοκή και συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της δικής σας κοινοβουλευτική Επιτροπής. Αυτό με φέρνει στην τελική μου ακροτελεύτια παρατήρηση και ολοκληρώνω. Και ο κύριος Χαραγή και ο κύριος Μέντεθ Ντεβίγο έθεσαν το ερώτημα τι γίνεται σε σχέση με μια πιθανή ένταξη ή προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα γίνει σε σχέση με τα κράτη, κύρωση νέου και υπό τις συνθήκες Λισαβόνας ήδη υπάρχει υπό το άρθρο, αντίστοιχο άρθρο μια πρόβλεψη ώστε εσωτερική απόφαση ομόφωνα του Συμβουλίου θα πρέπει πρώτα να αφορά τις ε, συνταγματικές ε, παραδόσεις των εθνικών κρατών μελών και έτσι θα εμπλακεί και το Κοινοβούλιο και αυτό οδηγεί τα κράτη-μέλη και τα θέτει στην εικόνα και έτσι δεν θα υπάρχει ίσως ανάγκη στο διεθνές ε, νομικό επίπεδο τα κράτη-μέλη να χρειαστεί να επικυρώσουν ξεχωριστά αυτή τη σύμβαση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και ευχαριστώ τον εισηγητή ιδιαίτερα κύριο Χάουρεγγι για αυτή την πάρα πολύ καλή ενημέρωση των συναδέφων για ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ίσως ο συνάδελφος Χάουρεγγι τώρα μπορεί να αντιδράσει σε αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν και να ακούσουμε το συμπέρασμα <clears throat> αυτής της πρώτης ανταλλαγής απόψεων. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, αν είμαι σε θέση να μπορέσω να απαντήσω σε τόσο πολλές και τόσο, τόσο εξειδικευμένες ερωτήσεις και παρατηρήσεις που έγιναν από τόσο πολλούς συναδέλφους. Θα προσπαθήσω να το κάνω, όμως φυσικά πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε ευκαιρία να συνεχίσουμε να απαντάμε αυτά τα θέματα και να ασχολούμαστε με αυτά, να ασχοληθούμε με αυτά όταν θα εκπονηθεί το συγκεκριμένο έγγραφο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. να ξεκινήσω αντίστροφα για την εκτέλεση, για την ε, ένταξη και την εκτέλεση των, νομολογιών. Νομίζω ότι είναι εκτελεστές οι νομολογίες, οι αποφάσεις του δικαστηρίου του Στρασβούργου και το ίδιο το δικαστήριο και το, ε, υπάρχει και το Συμβούλιο Υπουργών των Κρατών Μελών όσον αφορά τη σύμβαση που επομίζεται να ε, υλοποιεί τον έλεγχο όσον αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων του δικαστηρίου. Και είχαμε εδώ και πολύ πρόσφατα, και επιτρέψτε μου μια πολύ σύντομη αναφορά στην Ισπανία, υπήρξε ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα στην Ισπανία που απαγόρευε την πολιτική συμμετοχή των ομάδων, εκείνων των πολιτικών ομάδων που πρόσκυνται στην τρομοκρατία και το δικαίωμα σε σχέση με την ε, υποβολή υποψηφίων για τις εκλογές. Θεμελιώδες δικαίωμα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα για την Ισπανία. Και το δικαστήριο θεώρησε με θετικό πνεύμα αυτό το νομοθέτημα, αυτό το νόμο μια και σε σχέση με την ε, τρομοκρατία υπήρχε αυτή η απαγόρευση όσον αφορά κόμματα που επρόσκυντο στην τρομοκρατία. Αν δεν ήταν αυτή η νομολογία του ε, δικαστηρίου του Στρασβουργού να γνωρίζετε ότι θα ήταν υποχρεωμένη η Ισπανία να αλλάξει τον νόμο τον οποίο είχε εγκρίνει και να υπάρξει άλλο νομοθέτημα και εκεί να προβλέπεται το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής αυτών των ε, ε, ανθρώπων. Εδώ λοιπόν σε σχέση με την εκτέλεση λοιπόν και εφαρμογή της νομολογίας του Δικαστηρίου του Στρασβούργου δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία. Επίσης πρέπει να πούμε ότι πραγματικά βελτιώνεται και πολύ σωστά ερωτήθηκε πιο πριν αν πραγματικά δημιουργούμε ένα σύστημα αυθεντικής προστασίας που θα διασφαλίζει την ε, εφαρμογή και την εκτέλεση θεμελιωδών δικαιωμάτων όσο αφορά τους πολίτες. Ειλικρινά πιστεύω εγώ ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη σύμβαση συνεπάγεται πραγματικά μια νέα εγγύηση νομικής ασφάλειας και βεβαιότητας ότι αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως πολύ καλά είπαν διάφοροι συνάδελφοι δηλαδή την ίδια την ουσία ή την πεμπτουσία ή το ADN της ε, πολιτικής ε, παράδοσης και του πολιτισμού της πολιτικής μας παράδοσης είναι απόλυτα εφαρμοστά όλα αυτά τα δικαιώματα. Δηλαδή ένας πολίτης που για παράδειγμα <clears throat> σε σχέση με προσφυγή όσον αφορά το δικαστήριο του Στρασβούργου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται ή ένα νομοθέτημα ή όταν ένα κράτος μέλος εκτελεί κοινοτικό δίκαιο δεν μπορεί να προσφύγει στο, ε, ε, σήμερα δεν μπορεί να προσφύγει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δικαστήριο. Αύριο όμως ε, ναι. Και αυτό ως γεγονός μπορεί να επαρκέσει για να σκιαγραφίσουμε ότι ανοίγεται ένας πολύ μεγαλύτερος ορίζοντας, πολύ μεγαλύτερης νομικής ασφάλειας και βεβαιότητας. Και θα έλεγα ότι επιτυχάνουμε τον τετραγωνισμό του κύκλου, ας το πω έτσι, όσον αφορά την επίτευξη της ε, ε, διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών μέσω της επικύρωσης αυτής της σύμβασης. Και όσον αφορά το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο με την αρμοδιότητα που θα έχει και με δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, με όλα αυτά και ο κύριος Νταφ νομίζω τέλεια το εξέφρασε, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ένα δικαστήριο δεύτερο, ε, με συγχωρείτε, ε, επουσιώδες όσον αφορά το ΔΕΚ. Όχι, είναι ένα εξειδικευμένο δικαστήριο που ασκεί εξωτερικό έλεγχο όσον αφορά τις υποχρεώσεις, διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ασκεί αυτό τον έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση της σύμβασης. Δηλαδή, το δικαστήριο του Στρασβούργου έχει εξειδικευμένα αυτές τις αρμοδιότητες. Απλά και μόνο αυτές και επιμένω και εμένω σε αυτό και αυτό πρέπει να το αποσαφηνίσουμε απόλυτα. Τώρα, άλλες ερωτήσεις. Αν τα κράτη-μέλη θα μπορούν, θα είναι δυνατόν όσον αφορά άλλα μέλη της σύμβασης να ασκήσουν προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω σε σχέση με το άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, 33, 33 της σύμβασης μπορούν να το κάνουν αυτό πραγματικά, δηλαδή αποτελεσματικά, μπορεί ένα άλλο κράτο μέλο, ένα κράτο μέλο να ασκήσει προσφυγή κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, αναφερόμουν όταν είπα ότι δεν μπορούμε ο ένα να ασκήσει προσφυγή ή ε, αγωγή κατά του άλλου, αναφερόμουν αναμεταξύ μα στα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό μεταξύ κρατών μελών. Όμω, σε σχέση με ένα από τα ε, κράτη-μέλη ε, σε σχέση με ένα από τα κράτη της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, όταν υπάρχει μια παραβίαση όσο αυτό το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης ή της ελευθερίας των πολιτικών ελευθεριών αυτό το οποίο είπα στην αρχική μου εισαγωγή ότι σε σχέση με τις αρχές που εμπνέουν τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν πιστεύω ότι θα είναι δυνατόν και το λέω αυτό επειδή οι αρχές ε, για τη συνεργασία μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπουν να καταγγέλουμε ο ένας τον άλλον, το ένα κράτος μέλος ε, το άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει και αυτό να αποσαφινιστεί επίσης. Τώρα, συγγνώμη μια στιγμή να το βρω νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή, να υπάρξει καταγγελία σε σχέση με το δικαστήριο του Στρασβούργου, το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την ε, σχέση κάποιων ε, μελών με την ε, σύμβαση. Διότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη σύμβαση πρέπει να γίνει πάντα υπο, λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενη πρέπει να γίνει και με αυτό ε, υπό το πρωτόκολλο υπαριθμών 8 της ε, σύμβασης πρέπει να γίνει σεβόμενη τους μηχανισμούς που είναι αναγκαίοι και που διασφαλίζουν ότι τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούν από τρίτα κράτη και οι ατομικές ε, δράσεις θα, που θα υποβάλλονται κατά των κρατών μελών, δηλαδή με άλλα λόγια η δυνατότητα προσχώρησης Ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να, γίνεται, να γίνει σεβόμενη τους όρους του πρωτοκόλου και ένα από τα συνεπαγόμενα του πρωτοκόλου είναι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει αυτή την αυτοεξαίρεση τριών χωρών από αυτή τη σύμβαση. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα όσον αφορά αυτό το θέμα, ότι είναι ένας από τους όρους ε, της εφαρμογής και υλοποίησης της σύμβασης αυτή η συγκεκριμένη πτυχή. Τώρα, για ένα νόμο ή νομοθέτημα μπορεί να μην είναι συμβατός ένας νόμος με τις αρχές της σύμβασης και μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά εναντίον ενός νόμου ή εναντίον ε, της ε, τοποθέτησης ενός θεσμικού οργάνου. Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο δικαστήριο σε σχέση με τις ε, υποχρεώσεις που απορρέουν και που επιβάλλονται της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλους που έχει επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Και σε σχέση τώρα με τις χώρες, δεν ξέρω αν απάντησα επαρκώς και ακριβώς στις ανησυχίες σας για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω όμως οπωσδήποτε να σας πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι μέλος αυτής της σύμβασης και συμμετέχει πλήρως, με πλήρη δικαιώματα και δικαιοδοσία στο δικαστήριο και Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τροποποίηση του status quo για το Ηνωμένο Βασίλειο που ως μέλος της Σύμβασης ε, και του Δικαστηρίου αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ε, αυτό, ως μέλος, ε, επομίζεται τις υποχρεώσεις και τα όσα συνεπάγονται από αυτή την προσχώρηση. Τώρα, για το 14 νομίζω ότι τίθενται εδώ κάποιες ενστάσεις που, τις οποίες κατανοώ βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να εκινήσουμε από το εξής ο δικαστής ως μέλος ενός κράτους αποτελεί μέρος αυτού του δικαστηρίου και έχει δικαιώματα αλλά και περιορισμούς. Έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη συζήτηση μιας υπόθεσης που αφορά τη χώρα του αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει, δεν μπορεί να έχει ψήφο. Αυτό είναι ένας κανόνας της ίδιας της σύμβασης. Και αυτό εμπνέεται από τη λογική ότι όταν εξετάζει το δικαστήριο μια νομοθετική πράξη, ένα νόμο μια συγκεκριμένη χώρα, πρέπει ακριβώς ε, να εξετάζεται ποια είναι η ιδεοντολογική εφαρμογή και η ουσία αυτού του νόμου. Εισακούγεται λοιπόν ο δικαστής αυτού του κράτους, η άποψή του, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει. Δηλαδή η ανεξαρτησία του δικαστηρίου σε σχέση με την τοποθέτηση ενός ε, κράτους ε, γίνεται μέσω της έμεσης παρέμβασης ενός δικαστού που εξετάζοντας ε, ένα νόμο ή μια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη συγκεκριμένη εφαρμογή όσον αφορά συγκεκριμένο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δικαστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί, θα συμμετέχει, θα συμμετάσχει στην επεξήγηση των διατάξεων αυτού του νομοθετήματος που είναι υπό εξέταση για να δούμε αν παραβιάζει τις αρχές των θεμελιωδών ελευθεριών ή των ε, ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και μετά θα είναι το σώμα των δικαστών που θα λάβει την απόφαση χωρίς να επιτρέπεται στον Ευρωπαίο δικαστή να συμμετάσχει και να εκφράσει την άποψή του με ψήφο, ψηφίζοντας. Και αυτά λοιπόν νομίζω ότι μας οδηγούν στο να καταστήσουμε σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το είπα πιο πριν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι η ίστατη, ας το πω έτσι, αρχή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συμμετέχει όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε περίπτωση παραβίασής τους ή παράβασής τους και όσον αφορά και την εφαρμογή του δικαίου όσον αφορά τη σύμβαση. Έτσι το δικαστήριο, το αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή το 10, το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, θα εξετάζει σε σχέση με την εφαρμογή της χάρτας τα σχετικά, αλλά μόνο αν κάποιος ερμηνεύσει και πει ότι ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις θεμελιώδεις ελευθερίες που εντάσσονται και συμπεριλαμβάνονται στη χάρτα, στη σύμβαση, τότε θα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκείνο θα είναι αρμόδιο να εξετάσει και να κρίνει. Και εδώ δεν υπάρχουν ε, ε, τριβές ή ε, θέματα μη συμβατότητας μεταξύ της σύμβασης και της εφαρμογής της. Αναφέρονται αυτά τα θέματα και πρέπει να ερμηνεύονται ως εξής. Το δικαστήριο και η νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκείνο το οποίο πιθανότατα θα κάνει είναι θα προσανατολίζεται και θα εμπνέεται για τη συγκεκριμένη εφαρμογή των δικαιωμάτων που περιέχονται στη χάρτα και έτσι θα δρά ως ίστατη πηγή πρωτογενούς δικαίου όσον αφορά την εφαρμογή της ε, χάρτας ε, θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Δεν ξέρω αν χρειάζεται επίσης εδώ να προσθέσουμε και να πούμε και στον Πρόεδρο θα ήθελα με κάθε κατανόηση και συμπάθεια να πω ότι ίσως εδώ δεν υπήρξε η σωστή τοποθέτηση. Μέρος της αρχής για το ότι συμμετέχουμε θα προσχωρήσουμε σε αυτή τη σύμβαση σαφές είναι ότι δεν πρόκειται για προσχώρηση στο συγκοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκείνο το οποίο ε, είναι το περίπλοκο είναι το θέμα της συμμετοχής στην εκλογή των δικαστών χωρίς να συμμετέχουμε άμεσα στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και εγώ ίδιος όπως και άλλοι ε, συμμετείχα και εγώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο παρελθόν και θυμούμε πως ε, ψήφιζαν και τοποθετούντο και τι γινόταν με τους δικαστές ε, και σε σχέση με τους όσους προσέρχονται στις κάλπες εκλέγουν. Τώρα το θέμα είναι σε σχέση με τους τρεις δικαστές που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το αξίωμα του Ευρωπαίου Δικαστή πώς θα μπορεί να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Φυσικά όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα συμμετέχει στο, στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, σαφές. Νομίζω επίσης ε, είναι ορθό και αληθεύει ότι αν εγκριθεί το πρωτόκολλο υπαριθμό 14 πιθανότατο είναι ότι στις διαπραγματεύσεις που θα κάνουμε και θα γίνουν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με το Συμβούλιο της Ευρώπης διορθώνει ο μιλητής, θα μας οδηγήσει σε μια ανακαίνιση, καινοτομία, μεταρρύθμιση του ιδίου του Συμβουλίου δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει να υπάρξει εκπόνηση άλλου πρωτοκόλου, αλλά η αναζήτηση της ευελιξίας από πλευράς ε, δικαστικού σώματος σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αν θεωρεί ότι αυτό επαρκεί σε περίπτωση επικύρωσης από την ε, Ανώτατη Βουλή στη Ρωσία. Τώρα, αυτή η σύμβαση με όλες ε, τις ιδιομορφίες που έχει και μένω σε αυτό. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε υπογράψει τα κράτη-μέλη κάποια πρωτόκολλα. Όχι όλα. Και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο, όπως καλά είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, μιας προηγούμενης εξέτασης από τα κράτη-μέλη, τα οποία σε σχέση με την προσχώρηση δεν θα την εγκρίνουν αν δεν εξεταστεί υπό ποιου όρου θα γίνει η προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με ποια πρωτόκολλα. Φοβάμαι ότι αυτό θα διαρκέσει αρκετό χρόνο. Θα είναι μια περίπλοκη διαπραγμάτευση και διαβούλευση. Όμω πρέπει να γίνει αυτό προφανώ, διότι απαιτεί, απαιτεί κατηγορηματικά η συνθήκη τη Λισαβόνα και πρέπει να είναι σεβαστός ο τρόπος με τον οποίο έγινε και προβλέφθηκε η προσχώρηση των χωρών όσον αφορά την σύμβαση και πρέπει να είναι σεβαστά επίσης τα όρια τα οποία πάλι όπως αναφέρθηκε μη δημιουργίας νέων αρμοδιοτήτων και το πρωτόκολλο 8 ή το αντίστοιχο άρθρο της συνθήκης Λισαβόνας προβλέπουν ότι η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη σύμβαση δεν πρέπει να αλλοιώνει ή να έχει επιπτώσεις στην τοποθέτηση των κρατών μελών και σε σχέση με τα πρωτόκολλα που έχουν επικυρωθεί. Έτσι λοιπόν σε σχέση με πιθανές ε, εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις που ε, θα έχουν διατυπωθεί από τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα αυτές οι επιφυλάξεις ή εξαιρέσεις, να μην υπάρξει δηλαδή σε σχέση με την νομική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οποιαδήποτε αλλίωση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλες τις παρεμβάσεις. Σίγουρα δεν το κατάφερα να απαντήσω όλες τις παρεμβάσεις σας. Αλλά έχουμε επαρκή θέματα και νομίζω επαρκή χρόνο ε, καλύψαμε ασχολούμενοι με αυτά. Όταν θα υποβληθεί το τελικό έγγραφο, ας το πω έτσι, η πρώτη, το πρώτο σχέδιο της έκθεσης μου θα έχουμε την δυνατότητα να εξειδικεύσουμε πιο εξειδικευμένα σε μεγαλύτερο βάθος όλα αυτά τα θέματα. Θα λάβουμε υπόψη τις παρεμβάσεις και θα συνταθεί ε, το έγγραφο ακολουθώντας τις δικές σας συστάσεις και υποδείξεις. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα τώρα είναι ο χρόνος. Αλλά πριν να δώσουμε ημερομηνίε, θα δώσω το λόγο και πάλι στον Μέντε Δεβίγο. Για να μην αφήσουμε εκρεμές μετέωρο ένα θέμα από τη συζήτηση, θα ήθελα να το αποσαφηνίσω αυτό δεν υφίσταται opt-out, αυτοεξαίρεση τριών κρατών μελών στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει τέτοιο opt-out. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εφαρμόζεται στα 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο υφίσταται για τρία κράτη-μέλη, υφίσταται μία αναφορά στην εφαρμογή που κάνουν ή στην ερμηνεία που κάνουν σε σχέση με τα εθνικά δικαστήρια για αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει αυτοεξαίρεση για τη χάρτα αυτή. Η χάρτα αυτή εφαρμόζεται και στα 27 κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα το πρόβλημα είναι αυτό του χρονοδιαγράμματος. Γιατί όπως υποσχέθηκα, πρόθεσή μας είναι να επηρεάσουμε την παρέμβαση της Κομισιόν προς το Συμβουλίο, αλλά πρέπει να βιαστούμε. Και θέλουμε να κάνουμε και την ακρόαση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί με τους συντονιστές να, ποιον, να δούμε με τους συντονιστές ποιον και πότε θα ακούσουμε. Ε, αν θέλουμε να, κάνουμε, να προλάβουμε θα πρέπει ε, η έκθεση αυτή να ψηφιστεί μέχρι τις 7 Απριλίου. Θα τα καταφέρουμε. 7 Απριλίου, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διοργανώσουμε την ακρόαση για τις 17 Μαρτίου. 17 Μαρτίου ακρόαση και τελική ψηφοφορία 7 Απριλίου. Ένα έγγραφο το οποίο θα μπορεί να τροποποιηθεί, ένα γραπτό κείμενο πάνω στο οποίο να μπορούμε να εργαστούμε για τις 22 Φεβρουαρίου. Είναι στενά τα χρονικά όρια, αλλά είναι αναπόφευκτο αυτό αν θέλουμε να μπορέσουμε να παρέμβουμε αγκαίρω. Ο εισηγητή συμφωνεί. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν θα τα καταφέρουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5 της ημερήσια διάταξη. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την, ε, σε σχέση με τις λεπτομερείς διατάξεις άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μάρτιν έχει αναλάβει. Εδώ. Ναι, εδώ είστε. Α, δεν σας είχα δει. Λοιπόν, δώσω αμέσω το λόγο να μας κάνει την ε, εισήγησή του χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το καλό με αυτό το θέμα είναι ότι είναι πολύ λιγότερο περίπλοκο από το προηγούμενο και το να φτάσουμε σε συνένεση στην Επιτροπή θα πρέπει να είναι σχετικά εύκολο. Το σημαντικό πρόβλημα θα είναι, όπως και με το προηγούμενο, να συμφωνήσουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα. Αλλά να σας ε, εκθέσω πρώτα το ιστορικό για όσους δεν παρακολούθησαν την υπόθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρχήν είχε το δικαίωμα να δημιουργεί προσωρινές επιτροπές ε, έρευνας μέσω της συνθήκη του Μάστριχτ και αυτό για να διερευνήσει ισχυρισμούς για παραβιάσεις ή κακοδιαχείριση στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Η συνθήκη του Μάστριχ και τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας δεν δίνει λεπτομέρειες για το πώς θα πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι επιτροπές έρευνες, πώς θα λειτουργήσουμε με βάση ποιους κανόνες και ούτω καθεξής. Αυτό ανατίθεται σε μία, μάλλον ρυθμίζεται μέσω μιας διαθεσμικής διοργανικής συμφωνίας. Για να σας δείξω πόσο δύσκολο θα είναι θα δείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε να εργάζεται πάνω σε αυτό το 1992 αμέσως ε, με την συνθήκη της ε, του Μάστρα. Είχαμε δύο εκθέσεις ε, το 1995 ώστε να υιοθετηθούν οι κανόνες και ε, δεν θα με εξέπλησε να έχουμε ακόμα τρία χρόνια μέχρι ότου υιοθετηθούν οι νέοι κανόνες. Το κείμενο που υιοθετήθηκε τότε το 1995 είναι στους φακέλους σας δυστυχώς μόνο σε 11 γλώσσες διότι ε, τότε 11 γλώσσες είχαμε και μετά από την ε, δημιουργία διαφόρων επιτροπών έρευνας. Ε, προσέχαμε πολύ για να το χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα αυτό. Μόνο τρεις ερευνητικές επιτροπές έχουν ε, συσταθεί. Η πρώτη ήταν ε, για το καθεστώς διέλευσης, το δεύτερο για την τρελή αγελάδα και η τρίτη για την κρίση με τις ασφαλίσεις ζωής. Πολλοί ανησυχούν για τις αρμοδιότητες και για τις δυνατότητε των ερευνητικών αυτών επιτροπών να διεξάγουν το έργο τους. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες οι αρμοδιότητες μιας τέτοιας επιτροπής. Εγώ δεν πιστεύω πως πλέον συμφωνούν, συνάδουν με το πολιτικό κύρος αυτού του θεσμικού οργάνου. Ε, Το πρόβλημα που είχαμε αντιμετωπίσει ήταν ε, ότι δεν είχαμε πάντα πρόσβαση στα κείμενα, δεν μπορούσαμε να καλέσουμε μάρτυρες. Ε, και σε ορισμένε περιπτώσει ήταν αδύνατον να επιτευχθεί συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Επίσης, Αυτή η Επιτροπή οδήγησε στη δημιουργία ειδικών ερευνητικών επιτροπών και στα εθνικά κοινοβούλια. Και εκεί συμπεράναμε πω τα εθνικά κοινοβούλια είναι σε πολύ καλύτερη θέση ώστε να προβούν σε τέτοιε ερεύνε από ότι εμεί. Στην Ολομέλεια το 1997 υιοθετήσαμε μια έκθεση που ζητούσε από την διάσκεψη των Προέδρων να αναθεωρήσει τους κανόνες λειτουργίας των ερευνητικών επιτροπών. Και γιατί το κάνουμε τώρα, γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας αλλάζει τη διαδικασία για τις προδιαγραφές. Είναι το άρθρο 226 και αλλάζει το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει για τι λεπτομέρειε σύμφωνα με μια ειδική νομοθετική διαδικασία που θα έχει τη συγκατάθεση του Συμβουλίου και τη ε, Κομισιόν. Δηλαδή, η διαφορά είναι ότι εμεί έχουμε τώρα δικαίωμα πρωτοβουλία, ενώ παλιότερα έπρεπε εμεί να, να αναζητήσουμε τη συμφωνία των δύο άλλων θεσμικών οργάνων. Το καλό νέο είναι λοιπόν ότι έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλία. Το κακά νέο είναι ότι χρειαζόμαστε ακόμα τη συγκατάθεση Συμβουλίου και Επιτροπής. Ε, επίσης ε, ε, προχωρούμε με αυτό αυτή τη στιγμή γιατί οι αρμοδιότητες του Ombudsman είναι πέρα από τις αρμοδιότητε τη δική μα ερευνητική επιτροπή. Ο, ο, ο Ombudsman έχει πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες, μπορεί να έχει πρόσβαση στην ε, ε, στα έγγραφα, μπορεί να κλητεύει μάρτυρες και δεν είναι σωστό εμείς να έχουμε λιγότερες αρμοδιότητες από ότι ο Ombudsman. Η διαδικασία, Πρόεδρε. Επειδή τώρα η συνθήκη μας δίνει το δικαίωμα πρωτοβουλίας, προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα 41 του καταστατικού μας που είναι ο, εκείνος ο κανονισμός που καλύπτει το δικαίωμα πρωτοβουλίας που έχει το Κοινοβούλιο και απορρέει από τις συνθήκες. Εγώ προτείνω, επειδή έχει αλλάξει η διαδικασία, δεν θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον ισχύοντα κανόνα, αλλά να δημιουργήσουμε ένα νέο κείμενο τελείω. Αυτό βέβαια δεν μα εμποδίζει να βασιστούμε στους του κανόνε, αλλά να λειτουργήσουμε σαν να μεταρρυθμίζουμε ολόκληρο το κανόνα, μάλλον σαν να φτιάχνουμε νέο κανόνα, κανονισμό, παρά να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε τις ισχύουσες νομοθεσίες και θα πρότεινα να το κάνουμε σε δύο φάσει. Καταρχήν, και βεβαίω το λέω να γίνει σε δύο βάσει γιατί όπω σα είπα χρειάζεται συγκατάθεση των άλλων θεσμικών οργάνων. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μια ανέκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να την υποβάλουμε στα άλλα θεσμικά όργανα και να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις μαζί τους και έπειτα να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην ε, συμφωνία ώστε να έχουμε μια τελική έκθεση που θα φτάσει στην Ολομέλεια και θα εκθέτει τους νέους κανόνες. Εγώ νομίζω πως υπάρχουν τρεις τομείς όπου πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή όσον αφορά τη βελτίωση των κανόνων. Καταρχήν πρόσβαση στα έγγραφα. Και όπως ήδη αναφέρθηκα σε αυτό, το, ευκολότερο είναι να πούμε ότι η, μια ερευνητική επιτροπή θα πρέπει να έχει ακριβώ τα ίδια δικαιώματα όπω και ο Ombudsman όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα. Δεύτερον, θα πρέπει να βελτιώσουμε τα δικαιώματά μα όσον αφορά την κρίτευση μαρτύρων και φυσικά θα θα δεσμεύονται στο να απαντήσουν σαφώς τις ερωτήσεις μας και αναφέρω αυτή τη φράση διότι η έρευνα ε, η τελευταία απέδειξε ότι ορισμένοι από τους μάρτυρες δεν ήταν ε, πρόθυμοι να, απαντήσουν ε, στα ερωτήματά μας. Και έπειτα, ερευνητικέ μας ε, αρμοδιότητες θα πρέπει να διευρυνθούν και να έχουμε το δικαίωμα να, να ζητήσουμε τη βοήθεια του Εθνικού Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας. Θα πρέπει να τονίσω σαφώς και θα πρέπει να το κατανοήσετε πως εγώ δεν προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η ερευνητική μας επιτροπή να λειτουργήσουν σαν δικαστήρια δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ποινέ σε πολίτε κτλ. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η εθνική νομοθεσία όσον αφορά τη δική μα επιτροπή θα διαφέρουν ε, σε μεγάλο βαθμό, αλλά πιστεύω πω θα πρέπει ωστόσο να έχουμε το δικαίωμα για πλήρη πρόσβαση στην ενημέρωση. Και αυτό σημαίνει τόσο όσον αφορά τα έγγραφα, το προσωπικό που ασχολείται με αυτά και δικαίωμα έρευνα εν γέννη. Αυτό είναι ο στόχος. Προσπαθούμε να φτιάξουμε νέο κανονισμό και το χρονοδιάγραμμα είναι να σας φτιάξω εγώ μια γραπτή έκθεση για τη συνεδρίασή μα στις 17 Μαρτίου και 18 Μαρτίου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι στην Ολομέλεια πριν διακόψουμε για το καλοκαίρι και να μπούμε σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν μετά το καλοκαίρι. Ελπίζω, δεδομένε νέες σχέσεις με την Κομισιόν, ότι η Κομισιόν δεν θα δημιουργήσει πολλέ δυσκολίε, αλλά ειλικρινά σα λέω, προβλέπω πολλές σκληρέ διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ε, Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο να πάρει το λόγο. Ωραία. Θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό στις 17 και 18, είπατε, 17 Μαρτίου. Ναι, θα μας παρουσιάσετε μία έκθεση γραπτός στις 17 Μαρτίου. Εντάξει. Αυτό αποφασίσαμε λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο ε, θέμα, την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εδώ έχουμε τέσσερα σημεία στη μερίσια διάταξη, τέσσερις εκθέσεις που αφορούν τέσσερις νομοθετικές προτάσεις για να εποπτεύουμε καλύτερα την εξέλιξη των χρηματαγορών. Ε, η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Όμως η δημιουργία αυτών των τεσσάρων οργανισμών εποπτείας έχει επιπτώσεις θεσμικού χαρακτήρα. Γι' αυτό ασχολούμαστε και εμείς ε, με γνωμοδότηση προφανώς. Οι εκθέσεις είναι τέσσερις, αλλά επειδή μοιάζουν πάρα πολύ, γι' αυτό διορίσαμε ένα και μόνο εισηγητή, τον κύριο Μέντες Δεβίγκο. Τον παρακαλούμε λοιπόν τώρα να μας παρουσιάσει το θέμα το θέμα που αφορά την αυτονομία, την πολιτική ευθύνη των ε, εποπτικών αυτών αρχών, καθώς και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους και τη συμβατότητα με διάφορα συγκεκριμένα σημεία των συνθήκων. Ο κύριος Μέντες Δεβίκο έχει το λόγο. Σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζοντας αυτή την κοινοβουλευτική θητεία, ένας ε, καλός μου φίλος έλεγε ότι πιθανότατα η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είχε πάρα πολύ δουλειά στην έναρξη αυτής της θητείας. Μέσα και ο κύριος πολιτικός μας στόχος η συνταγματική χάτα και η συνθήκη είχαν επιτευχθεί. Νομίζω λάθος είχε κάνει, διότι η συζήτηση απόψε το αποδεικνύει. Πρώτον, σε σχέση και με την πρώτη αυτή συζήτηση για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το, Χάρτα Δικαιωμάτων. Τώρα ξεκινά λοιπόν αυτή η δουλειά, διότι οι θεσμικές πτυχές του νέου συστήματος ε, όσον αφορά τους ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα θεσμικό, σε βάθο ε, πολιτικό και νομικό που έχει επιπτώσεις ε, στα οικονομικά θεσμικά όργανα, οικονομικά, χρηματοοικονομικά, χρηματοπιστωτικά όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο και η πρώτη αναγνώρισή μου πρέπει να είναι προς αυτή την, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή που με διόρισε εισηγητή σε σχέση με την άποψη να δημιουργηθεί ένας εισηγητής ε, για κάθε μια θεσμική πτυχή που αναγνωρίστηκε ότι δεν θα ήταν το πιο όρθο. Διότι οι αρχές, ιδιαίτερα οι μικροαρχές, είναι ουσιαστικά οι ίδιες. Το να έχουμε λοιπόν διαφορετικούς ε, εισηγητές δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα οι διαφορετικούς συντάκτες γνωμοδότησης. Αυτό είναι μέρος ε, των θεμάτων που καλύπτονται και όπως πολύ καλά είπατε είναι η Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Θεμάτων η αρμόδια της ουσίας και που έχει διορίσει πέντε εισηγητές αν θυμάμαι σωστά δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Χρηματοπιστωτική Αρχή Γκαρθία Μαργάλιο για την μακροεποπτεία ε, και τον κύριο Κίγκολτ για την Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών και διαφορετικός εισηγητής όσον αφορά τις, την πτυχή των ασφαλιών. Έχουμε λοιπόν πέντε συνιστώσεις όσον αφορά τις προτάσεις αυτές που υπευλήθησαν το Σεπτέμβριο 2009 σαν συνέπεια ακριβώς και σαν απάντηση, αντίδραση στην χρηματοοικονομική κρίση και δεδομένη της ανάγκης να αποφύγουμε αυτό το οποίο είχε τότε παρουσιαστεί και είχε δημιουργηθεί κατά το παρελθόν, να μην επαναληφθεί κατ' στο μέλλον δηλαδή. Και υπάρχει βούληση, πολιτική, σαφής πολιτική βούληση να αφήσουμε πίσω πια μια ε, τέτοια φάση όπου ε, η επιτήρηση των χρηματοοικονομικών αγορών ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών κρατών μελών και οργάνων τους και η υπερεθνική εποπτεία βασιζόταν σε αρχές καλής πρακτικής, benchmarking ή ε, μέθοδο ανοιχτού συντονισμού κτλ. Όλα αυτά δεν λειτουργήσαν όμως ε, δυστυχώς και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο προώθησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό την Προεδρία και ιδιαίτερα υπό την Προεδρία του κυρίου Σαρκοζή προωθήθηκε το θέμα νομοθέτησης, νομοθετικής ρύθμισης αυτών των θεμάτων. Νομοθετικού έργου, νομο, νομοθετικού έργου που μεταφράστηκε σε τέσσερις κανονισμούς όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Συμβούλιο. Τέσσερις λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την σωστή ορολογία. Ήταν λοιπόν τέσσερα νομοθετήματα και μία απόφαση του Συμβουλίου που ε, υποβάλλεται στη σύμφωνη γνώμη και έγκριση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να αντιδράσουμε και να απαντήσουμε στη χρηματοοικονομική κρίση και να θεσπίσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας και επιτήρησης για τα χρηματοπιστωτικά θέματα. Αυτό είναι ο κύριος άξονας. Λοιπόν, καλώς. Τούτων λεχθέντων υπάρχει ένα θέμα που είναι αντικείμενο, όπως προανέφερα, απόφασης, όχι κανονισμού, αλλά απόφασης. Και είναι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων αφενός. Και αφετέρου έχουμε και τη δημιουργία μιας μακροοικονομικής χρηματοοικονομικής εποπτείας καθώς επίσης και μικροοικονομικών εποπτικών αρμοδιοτήτων. Κάνουμε λοιπόν λόγο και για τις συντάξεις και ασφαλιστικά θέματα και για τις άλλες συνιστώσεις. Θεώρησα πρόεδρε ότι ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσω το σύστημα PowerPoint διότι δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν όλα αυτά. Και ίσως έχοντας λοιπόν μια οθόνη όπου αυτά μπορούν να ανακεφαλαιωθούν και να τα δούμε ξεχωριστά καλύτερα. Εδώ κάνουμε λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων και για το Ευρωπαϊκό Σύστημα ε, Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας ή Επιτήρησης και βλέπετε ότι υπάρχει διπλή κατεύθυνση. Υπάρχουν εθνικές αρχές ε, εποπτείας χρηματοπιστωτικών θεμάτων που υφίστανται αυτή τη στιγμή και μένω και επιμένω το πρώτο σημαντικό στοιχείο θα συνεχίσουν να έχουν πρωτο, πρωταρχικό ρόλο και χαρακτήρα μέσα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η αρχική ας το πω έτσι προέλευση και αρχική δράση ήταν στο επίπεδο το εθνικό αρμοδιότητα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που δημιουργείται τώρα και είναι καινοτομία είναι οι ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας. Αυτό είναι το καινούριο. Και εδώ έχουμε τις τρεις αυτές τις οποίες προαναφέρθηκα. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο κάνουν και κάνει αυτές τις ευρωπαϊκές αρχές ε, χρηματοπιστωτικής επιτήρησης ε, και τι, πώς αντικαθιστούν τις ήδη οι φυστάμενες επιτροπές. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι και έχουμε την εκπόνηση τεχνικών ε, διατάξεων, technical standards. Εποπτεύουν ε, και ε, επιτηρούν για τη σωστή εφαρμογή του κοινοτικού νομικού πλαισίου μεριμνούν για την επίλυση τριβών και προβλημάτων που δημιουργούνται και παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις κατεπίγουσες. <clears throat> Έχουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο μέσα ακριβώς στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών που δίνονται σε αυτή την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή Υπηρεσία Εποπτείας έχουμε πρώτα τα technical standards, τεχνικές διατάξεις ε, και ρήτρε ε, που υποχρεωτικά θα πρέπει να διαβουλεύονται δημόσια Δηλαδή, θα πρέπει ουσιαστικά να διαβουλεύονται με τους αρμόδιους τομείς, επιχειρήσεις, στον χρηματοοικονομικό τομέα για παράδειγμα μετά από αυτή την πρώτη φάση διαβουλεύσεων η Ευρωπαϊκή Αρχή υιοθετεί ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο νομολογίας ή τεχνικών διατάξεων. Αυτή η έγκριση όμως δεν είναι αρμοδιότητα της ίδιας αυτής της αρχής. Τυπικά και επίσημα αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση και αυτή είναι εκείνη η οποία έχει αυτή τη δικαιοδοσία. Τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχθεί την πρόταση που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Εποπτείας να υπάρξει πλήρης έγκριση. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα κανονισμό με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που θα δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τι θα γίνει όμως αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνεί με την πρόταση που υποβάλλει η, αρχή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας σε σχέση με τεχνικές διατάξεις. Ε, λοιπόν εδώ είναι το πράγμα που δεν είναι απόλυτα σαφές και εδώ υπάρχουν και οι πρώτες αμφιβολίες ε, που υφίστανται αν την εγκρίνει εν μέρη ή θέλει να την τροποποιήσει. Και έτσι λοιπόν θα ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτήρησης για τους λόγους που ε, οδηγούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσουν αυτές τις προτάσεις τη. Εδώ έχουμε λοιπόν ε, μια τέτοια περίπτωση που πρέπει να ξαναγυρίσουμε, να ξαναδούμε δηλαδή την ε, ολοκλήρωση αυτού του, αυτού του εγχειρήματος. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ κάνουμε λόγο για τις αποστολές, την αποστολή και τις αρμοδιότητες ε, των χρηματοπιστωτικών αρχών σε σχέση με την συνεκτική εφαρμογή και ε, σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Ποια ε, περίπτωση εξετάζουμε εδώ. Εδώ εξετάζουμε την εξή περίπτωση, όπου μια εθνική αρχή κάνει μια εφαρμογή εσφαλμένη του κοινοτικού δικαίου. Ε, τότε λοιπόν μπορεί να συμβεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας να πει στην Εθνική Αρχή ακούστε εφαρμόζεται λανθασμένα αυτές τις ε, ρήτρε και η Εθνική Αρχή να δεχθεί αυτή την σύσταση. Μπορεί όμως να μην δεχθεί αυτή τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας η Εθνική Αρχή και τότε θα μπορεί να υπάρξει μια σύσταση που θα απευθύνεται στην Εθνική Αρχή τότε μπορεί να τη δεχθεί η Εθνική Αρχή ή να μην την απορρίψει ή να μην τη δεχθεί. Τι θα συμβεί αν η Εθνική Αρχή δεν δεχθεί τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας. Ε, τότε θα έχουμε μία απόφαση. Μία απόφαση που θα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχετικό συναφές θέμα. Και εδώ φυσικά έχουμε και την δυνατότητα η Εθνική Αρχή να δεχτεί μια τέτοια, διαδικασία, μια τέτοια σύσταση, οπότε κλείνει η διαδικασία αυτή ή όχι. Ε, και τότε λοιπόν η ε, Ευρωπαϊκή Αρχή μπορεί, μπορεί να απευθύνει τέτοιου είδους αποφάσεις ε, ατομικά στους όσους εμπλέκονται στην χρηματοπιστωτική ε, αγορά. Παρεμβάσεις τώρα κατεπήγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 10. Εδώ κάνουμε λόγο λοιπόν για περίπτωση ε, σοβαρού κινδύνου απορρίθμισης ή αποσταθεροποίησης της χρηματοπιστωτικής λειτουργίας, τότε αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει μια απόφαση και να απευθύνει, να επιβάλλει μια τέτοια απόφαση, ε, να συστήσει μια τέτοια απόφαση ε, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας. Και να υπάρξουν ατομικές τέτοιες περιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων ή συστάσεων προς τις εθνικές αρχές. Τι θα γίνει τώρα και πάλι νέου, αν συνεχίσει ε, την, ε, ε, συμφωνήσει η εθνική αρχή, τότε δεν συμβεί τίποτα. Αν όμως ε, δεν συμφωνήσει, τότε μπορεί να λάβει αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας όσον αφορά συγκεκριμένους συμμετέχοντες παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Και εν τέλει, το τέταρτο στοιχείο που προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η επίλυση διαφορών που μπορούν να υπάρχουν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν έχουμε το θέμα συντονισμού για την λήψη κοινών ρυθμίσεων και διευθέτησης με κοινό τρόπο μεταξύ διαφορετικών αρχών. Σε αυτή την περίπτωση η ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας μπορεί να παράσχει επικουρικά ε, τη συνδρομή της και να υπάρξει και η θέσπιση μιας προθεσμίας ώστε οι εθνικές αρχές να μπορέσουν να συμφωνήσουν. Αν δεν υπάρξει συμφωνία εφόσον έχει εξαντληθεί αυτή η προθεσμία ε, σε αυτή, την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας μπορεί να λάβει μια απόφαση που θα μεταφέρεται και θα επιβάλλεται στις εθνικές αρχές. Αν δεν την ακολουθήσουν οι εθνικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας μπορεί να λάβει μια απόφαση που θα έχει επίπτωση και θα εφαρμόζεται στις ε, ε, αρχές που θα συμμετέχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές αυτό είναι ο στόχος να υπάρξει ένα πλαίσιο που θα εντάσσονται σε αυτό όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι περίπλοκα. Βρισκόμαστε μπροστά στη δημιουργία ενός συστήματος αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκού χαρακτήρα για το σύστημα εποπτείας που δημιουργεί πρώτα μία ολόκληρη αρχή ε, οργάνων εποπτείας και δημιουργεί στη συνέχεια διαδικασίες και διεργασίες που δίνουν τη δυνατότητα ώστε αυτή η εποπτεία να μπορεί να εφαρμόζεται και όσον αφορά τις εθνικέ αρχέ εποπτείας και το καθιστώ σαφέ εκείνε οι οποίε έχουν την αρχική αρμοδιότητα και πρωτογενή αρμοδιότητα και σε περίπτωση δυνατότητας ε, να ε, ε, επιβάλλονται στους όσους συμμετέχουν στην αγορά συγκεκριμένες διατάξεις. Αυτό είναι το πλαίσιο και γι' αυτό έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το γενικό πλαίσιο αυτό πρόταση ή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα, πολλά ερωτηματικά. Και έχοντας συντάξει αυτή την εισαγωγή, αυτή την παρουσίαση, που ε, ήταν ίσως ε, ε, υπερβολικά συνεκτική, υπερβολικά με συγχωρείτε σύντομη, εκεί όπου θα βρίσκεται η, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ποιο επίπεδο θα είναι ή σε περίπτωση τριβών και αντιπαραθέσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα επιλύονται τέτοιες ε, τριβές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της τι λέει. Αν υπάρξει τέτοια περίπτωση τριβής, εγώ η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επεξηγώ τους λόγους που με αναγκάζουν να λάβω μια διαφορετική απόφαση από εκείνη που συνιστά η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας. Προφανώς είναι, ε, είναι ότι πριτανεύει η άποψη τελικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, σε σχέση με την ε, δημοκρατική ευθύνη και υπευθυνότητα που πάντα ζητεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δρουν σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο, αυτό με οδηγεί, Πρόεδρε, να θέσω ένα ερώτημα. Ένα νομικό σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό όλων αυτών των ερωτηματικών και ερωτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας. Και επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση. Η συνθήκη Λισαβόνας εγκρίθηκε, επικυρώθηκε. Όμως η τελική ανάπτυξη και εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων σε πάρα πολλές ε, αποφάσεις ε, που αφήνουν ε, ας το πω έτσι ερωτηματικά και δεν υπάρχει ένα τελεσίδικο καθοριστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να εντάσσονται. Αυτές οι κατεντολήν αρμοδιότητες ή μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε άλλες ε, αρχές κάνουμε λόγο σε σχέση με το αντίστοιχο ε, άρθρο η κατεκτέλεση του 298 διότι προφανώς εξαρτάται από την απάντηση που θα δώσουμε το τι θα συμβεί. Και είναι σαφές πάντα ότι στη συμμετοχή των συνομοθετών και εκείνων που έχουν μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δικαιοδοσία και αρμοδιότητα έχουμε διαφορετικά πλαίσια. Εδώ θα έπρεπε να κάνουμε λόγο για μια αναδιάρθρωση ή μια, ας το πω έτσι, μια, ένα νέο πλαίσιο με κατεντολήν εκτέλεση αυτών ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνουμε λόγο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εποπτείας, ε, για τη λειτουργία της και τις αρμοδιότητές της ε, και εποπτικές αρχές χρηματοπιστωτικών πράξεων τεράστια σημασία για την ενιαία εσωτερική αγορά. Πώς θα διαφυλάξουμε την αναγκαία διαφάνεια ή την μη δημοσιότητα κάποιων ευαίσθητων στοιχείων που δεν θα πρέπει να διαχέονται και να αποκαλύπτονται. Και εν τέλει νομίζω ότι στο σύνολο, στο ευρύτερο σύνολο αυτών των ε, αρχών εποπτείας και επιτήρησης που δημιουργούμε είναι κάτι που εν τέλει πρέπει να διασφαλίσουμε πρόεδρε τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποια θα είναι δηλαδή η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποια θα είναι οι, ευθύνες, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώς θα επιμεριστούν αυτές οι αρμοδιότητες και σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή είναι μια ανταλλαγή απόψεων πρόεδρε που προβλέπεται από την ημερήσια διάταξή μας αυτό ήθελα να κάνω να επεξηγήσω και να τηρήσω και να περιοριστώ στα τέσσερα άρθρα τα οποία θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά. Υπάρχουν και άλλα τα οποία δημιουργούν όμως λιγότερες ε, αμφιβολίες όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Εποπτείας ε, ή των συστημικών προσπαθειών επιτήρησης. Όπως είπα αυτό αφορά την ίδια την αρμοδιότητα των αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Γι' αυτό ο εισηγητής σας εγώ, Πρόεδρε, θέλω να ακούσω τώρα, να φουγκραστώ τις απόψεις των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ώστε να μπορέσω να καταλήξω σε μια δυνατότητα εξειδίκευσης αυτών των στοιχείων που ε, εκπονούνται σήμερα και να υποβληθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ρυθμισή τους, γνωρίζοντας ότι οτιδήποτε κάνουμε εκείνο που θα πρέπει είναι να είναι λειτουργικό και να χρησιμοποιηθεί στο τέλος εποφελώς για κάτι. Πρέπει να το κάνουμε λοιπόν με σαφή συντονισμό την, με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Έχουμε λοιπόν εδώ θέματα τα οποία τίθενται στον χρηματοοικονομικό νομισματικό κόσμο και γίγνεσθε και πρέπει να βρούμε δυνατότητες με μεγαλύτερη διαφάνεια να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα και πρέπει να υπάρχει ένα νόημα και μια λογική εγγενής από πλευράς νομικής αυτών των ρυθμίσεων και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε πολύ στενά με τους πέντε εισηγητές από πλευράς της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μέντες Τεβίγκο. Οι εισηγητέ τη οικονομική και νομισματική επιτροπή είναι πέντε, αλλά εμεί έχουμε τέσσερι εκθέσει. Πώ γίνεται αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με τα νούμερα. Όχι πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν συμπεριλάβατε εσεί εδώ, σε αυτόν τον υπολογισμό. Α, έχει... Δεν έχει συμπεριληφθεί αυτό η μακροοικονομική εποπτεία και επιτήρηση. Εσείς έχετε ε, συνενώσει δύο πρόεδρε. Είναι τέσσερις, τέσσερις είναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είναι δύο των συστημικών κινδύνων και η άλλη είναι η εποπτεία, αλλά η, από πλευρά εισήγηση ε, ε, έχουμε πέντε θέματα με τέσσερις εισηγητές. Εντάξει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πώς παρουσιάσατε ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Μας κάνατε μια θαυμάσια παρουσίαση. Φυσικά κάτι πρέπει να διαβάσουμε κιόλα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια γνωμοδότηση πολύ σωστή, πολύ ικανοποιητική. Ο κύριος Μέσορ Σμιτ. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ καλή παρουσίαση και οπτική αλλά και επί της ουσίας από πλευρά σας. Μεγάλο μέρος του Σαββατοκύριακου το ανάλωσα διαβάζοντας αυτά για να έχω εξοικειωθεί κάπως πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θεματικό πλέγμα. Ευχαριστώ λοιπόν για την εισήγηση, την παρουσία σας. Θεωρώ όπως είπατε κύριε Μέντε Βίγκο ότι υπάρχει μια σειρά ερωτηματικών και θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν γενικά εκείνο το οποίο διαρωτώ με είναι για ποιο λόγο αυτά τα νέα όργανα δεν χαρακτηρίζονται ως ε, νομικού δικαίου ε, οργανισμοί ή υπηρεσίες. Είναι αποφασιστικού χαρακτήρα αυτού. αυτό. Αν θέλουμε να αποφύγουμε μια οικονομική κρίση στο μέλλον πρέπει ευθύς εξ αρχής να έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη, το δυνατόν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτά τα θεσμικά όργανα. Μέγιστη εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το σημείο καμπής για να ελπίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί μια τέτοια χρηματοοικονομική κρίση στο μέλλον. Και έχοντας εμπιστοσύνη ε, οι πολίτες σε αυτά τα νέα θεσμικά όργανα πρέπει να είναι και υπεύθυνα ταυτόχρονα αυτά τα όργανα και πρέπει να είναι σαφές ότι θα πρόκειται για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρεις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες. Μετά, για το θέμα του σε ποιο βαθμό ας το πω έτσι, οι προτάσεις, συστάσεις, υποδείξεις προς τις εθνικές αρχές εποπτείας ε, θα πρέπει να, είναι δημοσι... να δημοσιεύονται, να είναι δημόσιου χαρακτήρα και να διεξάγονται σε ένα ανοιχτό δημόσιο πλαίσιο. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι να υπάρχει δημοσιότητα εκτός αν είναι απόλυτα αναγκαίο να συμβαίνει το αντίθετο και να είναι κάποια πράγματα ε, να θεωρούνται θέματα εμπιστοσύνη. Γιατί για να υπάρξει εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις είναι αναγκαίο να υπάρχει δυνατότητα ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα. Φυσικά υπάρχουν θέματα εμπιστευτικού χαρακτήρα όσον αφορά την οικονομία. Ω σημείο κίνηση όμω, ω γενική αρχή, πρέπει να ισχύει η δημοσιότητα και ο δημόσιο χαρακτήρα ε, αυτών των δράσεων και τοποθετήσεων. Αυτό για τον δημόσιο χαρακτήρα αυτών των ε, διεργασιών. Μετά στη συνέχεια για την αναλογία, το συσχετισμό δυνάμεων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατικών αρχών και των κοινοτικών ε, θεσμικών οργάνων που δημιουργούνται με εποπτικές αρμοδιότητες. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα νέα θεσμικά όργανα να έχουν μια το δυνατόν ισχυρότερη εκκίνηση ή αφετηρία και να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους τα, οι εθνικές αρχές εποπτείας. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να πρέπει να παρακαλούν ή να οικετεύουν εθνικές αρχές για να τους διαβιβάζουν και να τους διαθέτουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Πρέπει λοιπόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτόματα να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν οι κρατικές ε, ε, ε, αρχές εποπτείας. Μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης. Και μετά όσον αφορά τις διατάξεις που αναφέρετε στη δική σας γνωμοδότηση και στην παρουσίασή σας, τι γίνεται εδώ η Εκτελεστική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Εκτελεστική Επιτροπή για την Εποπτεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται. Εντάξει, το θέμα είναι ποια δικαιώματα θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι απόλυτα φυσικό ότι δεν είναι μόνο το θέμα της ε, Αρχής Εποπτείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιμερίζονται αρμοδιότητες, αλλά και το όργανο που εκπροσωπεί τους πολίτες των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέκεται και αυτό. Στη χώρα μου δεν θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει, για παράδειγμα, αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο, πόσα αρχές φερεγγιότητας και ρευστότητας μπορούν ε, να αποτελέσουν αντικείμενο ε, εξέτασης ή διαβούλευσης χωρίς να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαβουλεύσεις και με το Συμβούλιο. Τώρα, και για τη διαδικασία συνδιαλλαγής ή ε, επίλυσης διαφορών σημαντικό θέμα αυτή η διαμεσολαβητική αρμοδιότητα. Να μπορεί να, διαμεσολαβ... να ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο αυτή η αρχή εποπτείας όταν υπάρχει ένα ε, θέμα τριβής μεταξύ δύο ε, κρατών μελών. Αυτό όμως μπορεί να είναι χρονοβόρο. Βλέπουμε πως κατέρευσαν μεγάλα θεσμικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσα σε μια εβδομάδα. Σαν χάρτινη πύργη. Δεν μπορούμε μια χρονοβόρο διαδικασία λοιπόν ε, να την χρησιμοποιήσουμε με αρχές στις οποίες θα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για να υπάρξει συνδιαλλαγή, διαμεσολάβηση μέσα σε χρονοβόρες διαδικασίες. Πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, με πολύ πιο γοργούς ρυθμούς. Έχω λοιπόν αμφιβολίες για αυτό το βραδύ ρυθμό. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Αρχή Διαμεσολάβησης και Επίλυσης Διαφορών για την πρέπει να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη κανείς σε αυτήν ότι πραγματικά θα μεριμνά ώστε οι αγορές να λειτουργούν σωστά όπως πρέπει. Best practices από τρίτες χώρες, βέλτιστες πρακτικές από την Ελβετία, της ΕΠΑ, την Κίνα για παράδειγμα πρέπει να αντλούνται ως ε, βάση το δυνατόν ευρύτερη για να μπορούμε να δράσουμε με τον καλύτερο, πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Και εν τέλει και κάτι άλλο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε το δυνατόν σαφέστεροι όσον αφορά διαδικασίες. Τις διαφανέστερες, σαφέστερες διαδικασίες με τους γοργότερους ρυθμούς και τη γοργότερη αλληλουχία για να είμαστε αποτελεσματικοί ώστε να είναι ανεξάρτητα τα όργανα από τα κράτη-μέλη. Το θεωρώ σωστό αυτό, να είναι ανεξάρτητα. Αλλά για τον τρόπο πώς θα ψηφίζουν, πώς θα δρούν αυτά τα θεσμικά όργανα, πρέπει να δούμε το, στο Συμβούλιο τι γίνεται. Δηλαδή πάλι έχουμε θέμα κρατών μελών και εδώ έχουμε το θέμα του μεγέθους των κρατών μελών και της επιρροής τους. Αφενός λέμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες από εθνικά συμφέροντα, από κρατικά συμφέροντα. Από την άλλη όμως πλευρά δεν θέλουμε να έχουμε μία ε, διεργασία όπου τα μεγάλα κράτη θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή σε σχέση με τα μικρότερα. Όταν θεωρεί κανείς για παράδειγμα ότι δεν θα πρέπει να διαδραματίζουν εθνικά συμφέροντα ε, ένα συγκεκριμένο ρόλο, τότε θα πρέπει να έχουν μία ψήφο τα κράτη, τα κράτη-μέλη. Μία ψήφο το ένα, μία το άλλο, άσχετα από μέγεθος, ώστε να μην επηρεάζει το μεγαλύτερο κράτος μέλος το μικρότερο. Σωστό είναι το πλαίσιο στο οποίο έχετε εκπονήσει τις προτάσεις σας, πολλά όμως πρέπει να γίνουν ακόμα. Μπορώ να σας διασφαλίσω βέβαια ότι και εγώ θα σας υποστηρίξω παρότι εκπροσωπώ μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, για την προσφορά σας να συνεργαστείτε. Ο κύριος Φερχόφσταντ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μέντε Στεβίγκο για αυτή την πρώτη έκθεσή του και θα ήθελα να του πω ότι κατά την άποψή μου είναι θετικό το να έχουμε ένα και μόνο εισηγητή για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τέσσερις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί αν έχουμε πολλούς, είναι πιο δύσκολη η συνομιλία. Με τέσσερις, ε, με τέσσερις ε, εισηγητές ε, θα συζητήσουμε τέσσερις φορές. Η Κομισιόν διάλεξε μια συγκεκριμένη διαδικασία για την πρότασή της και στην ΕΟΚΕ έχει, υπάρχουν τέσσερις ε, εισηγητέ, βέβαια. Οι προτάσεις της Κομισιόν υποβλήθηκαν στην ε, ΕΚΟΝ, στην Οικονομική Επιτροπή. Ε, οι προτάσεις είναι τέσσερις γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι νέες εποπτικές αρχές έχουν τέσσερις, αποτελούνται από τέσσερις πυλώνες. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση επί της ουσίας αυτών των προτάσεων τώρα. Κατά την άποψή μου, η ουσία θα πρέπει να συζητηθεί στο εσωτερικό της Οικονομικής Επιτροπής, η ουσία αυτών των προτάσεων. Γιατί εκεί είναι γνωστές οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις. Ε, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι στο εσωτερικό της ε, Επιτροπής ΕΚΟΝ υπάρχουν ε, νομομαθείς όπως και εδώ, αλλά πολλοί κόσμος είναι νομικός. Δεν ε, σπανίζει το είδος. Πριν μπούμε στα θεμικά, θεσμικά θέματα και στα νομικά θέματα της ε, πρότασης, θα ήθελα να σας πω ότι οι προτάσεις μοιάζουν να είναι πολύ καινοτόμε, ενώ δεν είναι τόσο πολύ καινοτόμε. Η Τρεις υπηρεσίες για την ε, μικροπροληπτική εποπτεία υπάρχουν. Επίσης, ε, η ομάδα Λαμφαλουσί δούλεψε πέρυσι και κατέληξε σε αυτές τις ε, υπηρεσίες. Έτσι δημιουργήθηκε η νομική αυτή πραγματικότητα που είναι οι, οι agencies. Η επιρροή της ομάδας Λαμφαλουσί ήταν μεγάλη. Είναι καλό αυτό. Πέρα από την μικροπροληπτική ας πούμε, διάσταση, υπάρχει και μία υπηρεσία, μία agency, η οποία θα πρέπει να αποφανθεί για τους συστημικούς κινδύνους των χρηματαγορών. Αυτό που δεν είναι επίσης καινούριο είναι ότι για τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις τράπεζες, τα ταμιευτήρια, ε, τις ασφάλειες οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες ακόμα και σήμερα όπως και στο παρελθόν. Όταν πρόκειται για διασυνοριακές δραστηριότητες έχουμε καμιά τριανταριά ή σαρανταριά τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω. Κάτι την άποψή μου ε, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερε τράπεζε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ο τραπεζικό τομέα είναι πιο σημαντικό. Υπάρχουν κάποια συνταξιδοτικά ταμεία, κάποια ταμιευτήρια επίση που είναι διασυνοριακά και που θα υπόκεινται σε, αυτή τη νέα μορφή εποπτείας. Θα ήθελα να προσθέσω ακόμα το εξή. Τελευταίο εισαγωγικό σημείο. Όλα αυτά δεν έχουν συζητηθεί ακόμα ε, στην ΕΚΟΝ ε, στους τέσσερις, ε, από τους τέσσερις εισηγητές που προέρχονται από τέσσερις διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Γιατί συζητούν αν αυτές οι προτάσεις πάνε αρκετά μακριά. Και υπάρχουν φήμε ότι κάποιοι εισηγητέ θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξε αυτέ οι προτάσεις. Πέρασε, ε, ξέρουμε ποια είναι η κρίση, ε, τώρα κάπως έχουμε προχωρήσει. Ακόμη και ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Μπαρόζο, αλλά το είπε και στο Κοινοβούλιο και εκτός Κοινοβουλίου. το Δεκέμβριο στο ΕΚΟΦΗΝ έγιναν κάποιες προτάσεις, ιδίως σε τρεις πτυχές της μικροπροληπτικής εποπτείας. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια έντονη προειδοποίηση ότι βασίζεται ο κ. Μπαρόζο στο Κοινοβούλιο για να καταστήσει πιο φιλόδοξη την πρότασή του. Επομένω, είναι λίγο παράδοξη η κατάσταση, κ. Μενδέστε Θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για την προ όφελο της ΕΚΟΝ, αλλά δεν ξέρουμε τι κατεύθυνση παίρνει η συζήτηση στο εσωτερικό τη ΕΚΟΝ. Νομίζω ότι οι τέσσερις εισηγητές που εμφανίζονται προς τα έξω με μία φωνή, στην πραγματικότητα έχουν επικρίνει ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξη αυτή η πρόταση. Πάνε πιο μακριά από τη σημερινή πρόταση. Εδώ ακριβώς μπορεί να παίξει ένα ρόλο η Επιτροπή μας, γιατί χάρη στις συστάσεις μας, οι τέσσερις συζητητές αυτοί και η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν, να παρουσιάσουν προτάσεις πιο φιλόδοξες από αυτές που έχουμε επιτάπητος. Πρέπει να δώσουμε μια θεσμική και νομική γνωμοδότηση. Αυτή η γνωμοδότηση πρέπει να μπορεί να βοηθήσει τους τέσσερις συζητητές της ε, ΕΚΟΝ για να φτάσουν σε ένα έγγραφο το οποίο θα είναι πιο φιλόδοξο από τις προτάσεις που έχουμε σήμερα. Τι είναι λοιπόν αυτός ο πιο φιλόδοξος, ποιος είναι αυτό ο πιο φιλόδοξος προσανατολισμός. Στο μέλλον στην Ευρώπη θα έχουμε 31 αρχές και φορείς που θα ασχολούνται με την χρηματοπιστωτική εποπτεία. 27 στο, σε εθνικό επίπεδο, ε, μία μακροπροληπτική και, τρι, ε, και τρεις μικροπροληπτικές. 31. Μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε μα ξεπέρνανε. 55 ή 60 φορεί έχουν. Υπάρχουν 50 ε, των ε, πολιτιών και υπάρχουν και κάποιες ε, αρχές εποπτικές ε, ομοσπονδιακές. Είναι 55 ή 65, 60 ή 65. εδώ κατά την άποψή μου και κατά την άποψη της ομάδας μου θα έπρεπε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της διατήρησης των εθνικών αρχών ε, που ασχολούνται με τις εθνικές ε, αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα ήταν να έχει μόνο μία εποπτική αρχή και όχι τέσσερις που θα ασχολούνταν και με την μικρό και με τη μακροπροληπτική εποπτεία. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη μικρο και μακροπροληπτική εποπτεία φυσικά. Η μακροπολιτική υποπτία επιτρέπει να καθορίσουμε τον συστημικό κίνδυνο, αλλά θα πρέπει να βασιστούμε σε πληροφορίες που προέρχονται από το προ, ε, μικροπροληπτικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα εδώ μοιάζει να σαν να αναπτύσσεται μία φούσκα γύρω από το χρηματοπιστωτικό τομέα. Όχι. Πρέπει, πρώτα να στηριχτούμε στο μικροπροληπτικό επίπεδο, μετά στο μακροπροληπτικό και να δούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο. Να δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες, ε, τα συνταξιδοτικά ταμεία και τις ασφάλειες. Οι τράπεζες, σημαντικότητα, είναι ανταγωνίστριες των συνταξιδοτικών ταμείων. Ε, αλλά και, και οι μεν και οι δε επενδύουν στο ίδιο προϊόν, προϊόν. Θα πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν και τις τράπεζες και τα συνταξιδοτικά ταμεία και τις ασφάλειες. Εγώ ανήκα στο μεγαλύτερο συνταξιδοτικό ταμείο της Ευρώπης. Είμαι αντιπρόεδρος ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο του και συνέχεια συνομιλώ με τράπεζες. Στο μέλλον θα ελέγξουμε αυτούς τους οργανισμούς με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε σαφέστατα την άποψή μας γιατί υπάρχουν από τη μία οι μικροπροληπτικές αρχές, οι οργανισμοί που ασχολούνται με τις ε, αγορές, με τις ε, τράπεζες, με τις, ε, τα στεξιωτικά ταμεία και τις ασφάλειες και θα πρέπει να έχουν νομικές ευθύνες. Θα πρέπει να έχουν λοιπόν μια νομική προσωπικότητα. Όμως στην πρόταση μπορεί να μειονεκτήσουν απέναντι στην Κομισιόν. Κοιτάξτε, ή θα έχουν μια πραγματική νομική προσωπικότητα και θα έχουν και την τελική απόφαση ή όχι. Αλλά εδώ δεν γίνεται έτσι. Η Κομισιόν τελικά μπορεί να κυριαρχήσει. Στα πλαίσια του μακροπροληπτικού ελέγχου που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή η agency, αυτός ο οργανισμός πάλι ξεπερνιέται από τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο πιο συγκεκριμένα όταν υπάρχουν δημοσιονομικές περιπτώσεις και όταν υπάρχει η απαραίτητη ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Ε, αυτό λοιπόν συνιστά πρόβλημα. Το θέμα είναι, πρέπει να δώσουμε όλες τις αρμοδιότητες στις υπηρεσίες για τον μακροπολιτικό και μικροπολιτικό έλεγχο και σε μία περίπτωση να είναι η Κομισιόν, σε άλλη περίπτωση τα κράτη-μέλη και τελικά το Συμβούλιο να αποφασίζουν εν τέλει όταν υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη. Και τελικά πρόκειται για δικές τους αρμοδιότητες που έτσι ξύνουμε. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Δεύτερον, η δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να πει ότι τίθεται ένα θέμα αποτελεσματικότητας εδώ. Έχουμε τρεις μικροπρονιακές, μικροπροληπτικές ε, υπηρεσίε, οργανισμούς. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα υπάρχει μια επιτροπή προφανώς από πάνω που θα συνεδριάζει για να διατητεύσει σε αυτές τις διαφορές. Επομένως, για τις ε, τράπεζες θα έχουμε μία υπηρεσία, μία για τις ε, ασφάλειες, άλλη για τις ασφάλειες. Θα υπάρχει και μία διευθύνουσα, ας πούμε, επιτροπή για τις ε, πάνω από αυτέ τι μικροϊπηρεσίε που θα αποφασίζει τελικά. Είναι αποτελεσματικό αυτό το σύστημα. Δεν νομίζω. Η Επιτροπή μα θα πρέπει να γνωμοδοτήσει με βάση τη νομική αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος. Γιατί να μην έχουμε μία και μόνη υπηρεσία, έναν οργανισμό με ένα τμήμα μακροπροληπτικό, ένα τμήμα μικροπροληπτικό και στο μικροπροληπτικό να έχουμε τα ταμεία, τις τράπεζες ε, και τις ασφάλειες. Υπάρχουν τρία οικονομικά κέντρα, το Παρίσι, η Φραγκφούρτη και το Λονδίνο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις τρεις αγορές. Θα πρέπει και αυτές κάπως να εκφραστούν μέσα από κάποιες υπηρεσίες, οργανισμούς. Εμείς ως συνταγματική υπηρεσία θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε ε, στην Οικονομική Επιτροπή και να της πούμε ότι δεν είναι αποτελεσματικός αυτός ο μηχανισμός. Θα πρέπει να έχουμε μία υπηρεσία με διαφορετικές γενικές διευθύνσεις ή διαφορετικά τμήματα που δουλεύουν μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Και το ίδιο για τον μακροπροληπτικό έλεγχο και εποπτεία. Θα ασχολείται αποκλειστικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία και θα συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή η agency, αυτός ο οργανισμός. Τέλος, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς μπορούμε να καθορίσουμε το ρόλο του στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει μια ετήσια έκθεση, όπως γίνεται και στα κράτη-μέλη μας. Μια έκθεση αυτών των ε, οργανισμών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι το ελάχιστο ελαχιστότατο που μπορεί να γίνει. Κάθε χρόνο δηλαδή θα πρέπει να γίνεται μια ετήσια αξιολόγηση του έργου που έχει γίνει από τους νέους αυτούς ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. ή μάλλον εποπτικούς οργανισμούς. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε δύο γνωμοδοτήσεις. Ή μάλλον, θα πρέπει να φασίσουμε για δύο πράγματα. Να έχουν νομική προσωπικότητα αυτοί οι οργανισμοί. Ή να λαμβάνονται αποφάσεις εν τέλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και το Συμβούλιο τελικά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και δεύτερο, δεύτερο θέμα. Να πούμε, δημιουργείται μια σειρά από οργανισμούς με ξεχωριστές νομικές προσωπικότητες και από πάνω είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε και ένα μηχανισμό διαιτησίας σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές απόψεων. Εμείς, ΑΦΚΟ, προτείνουμε σε εσά Συμβούλιο να έχετε μόνο μία αρχή εποπτείας οικονομικής, όπου θα εντάσσονται όλα αυτά τα στοιχεία ε, στα πλαίσια διαφορετικών γενικών διευθύνσεων, διαφορετικών τμήματων. Αυτά, ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Γεωργάκη. Μάλιστα. Να τα δούμε ένα προς ένα. Μετά από την παρέμβαση του κυρίου Φερχόφστα, θεωρώ κατάλαβα ότι έχουμε περισσότερα προβλήματα από όσα νομίζαμε. Γιατί αν προχωρήσουμε με μια πρόταση διοργανωτική διαφορετική από εκείνη που έχει προτείνει η ΕΚΟΝ και όπου προφανώς έχουν συμφωνήσει επ' αυτή τα μέλη της Επιτροπής δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα δεχθεί η δική μας άποψη πραγματικά να μην ξεπερνά αυτά τα πλαίσια που ήταν η πρόθεση της γνωμοδότησης από πλευρά μας. Παρότι μετά από τα όσα ανέφερε ο κύριος Φερχόφστατ, θεωρώ ότι είναι λογικά αυτά όμως αυτό με οδηγεί σε μια σκέψη ακόμα πιο περίπλοκη ως πρόβλημα. Να ερωτήσουμε δηλαδή, να διαρωτηθούμε αν πραγματικά η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καθορίσει αυτό το πρότυπό τους ε, της ε, παρέμβασης από πλευράς τους. Για όλο αυτό το νέο επίπεδο και πλαίσιο το οποίο απορρέει μετά τη χρηματοοικονομική κρίση για την εποπτεία, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών ε, συναλλαγών και πράξεων. Με άλλα λόγια, Έχω την εντύπωση ότι ακόμα η αρχιτεκτονική δομή, α το πω έτσι, η αρχιτεκτονική της δημόσιας παρέμβασης ή επέμβασης στα χρηματοπιστωτικά θέματα μετά την κρίση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν έχει δομηθεί ακόμα. Έχω ακόμα την εντύπωση ότι ακόμα βρισκόμαστε σε έναν αγώνα, σε μια προσπάθεια μέσα στην Ευρώπη και μέσα στην λέσχη G20 και στην συνάντηση του Ιουνίου του Καναδά κάτι θα πρέπει να αναφερθεί και γι' αυτό επίσης. Δηλαδή ποιες δομές θα θεσπιστούν για τον έλεγχο για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών, κάποιων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και φυσικά κάποιων χρηματοπιστωτικών οργάνων και θεσμών επίσης σε κάθε χώρα. Και πώς θα συντονίζονται όλα αυτά σε διεθνές επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και φοβούμε ότι ακόμα αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν διευθετηθεί. Παρακολουθούμε μια ενρευστό συζήτηση δηλαδή σε διαρκή εξέλιξη για φορολογικά θέματα, για χρηματοπιστωτικά θέματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για τοξικά ομόλογα, για για ε, μπόνους ομόλογα, χρεόγραφα και έχουμε νέα στοιχεία όσον αφορά τον, τους ελέγχους και την εποπτεία όσον αφορά τις ε, ε, χρηματοπιστωτικές δράσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι όλα αυτά ακόμα εκκρεμούν και πρέπει να καθοριστούν. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και τώρα, σε σχέση με το κριτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Οικονομικών Νομισματικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν τελεσίδικα ρυθμίσει όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό απλά και μόνο εφιστώ την προσοχή του εισηγητή στο πρόβλημα το ότι σε ένα μέρος των προτάσεων του Φερχόφστατ μα οδηγεί σε μια αντίστοιξη, σε μια διαφορετική τοποθέτηση ως προτύπου που δεν θα τη δεχθεί μάλλον η Επιτροπή ΕΚΟΝ όσον αφορά συνενέσεις και δική της αποδοχή και στο σημείο κατά πόσον αυτά μπορούν να γίνουν όλα αποδεκτά. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θέσω είναι κάπως το εξή. Ποια είναι η μορφή φύση αυτών των υπηρεσιών, των οργάνων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η παλαιά αντιπαράθεση γαλλογερμανική. Η Γερμανία θέλει μια ανεξάρτητη ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από πολιτικέ ε, μονάδε ή πολιτικέ πολιτική επέμβαση παρενέργειες και απομακρυσμένοι από τις πολιτικές παρεμβάσεις και έχουμε για παράδειγμα και την άλλη θέση της ε, ε, που θέλουν μια περισσότερη ε, επέμβαση πολιτική και παρέμβαση πολιτική της Ένωσης στα οικονομικά νομισματικά. Διαρωτώ τα όργανα τα οποία δημιουργούμε σε ποια τροχιά θα τεθούν και υπό ποια αρμοδιότητα θα βρίσκονται. Υπό την τροχιά και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των Ευρωπαϊκών Πολιτικών ε, ε, Θεσμών. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να έχουμε ένα σύστημα κοινοβουλευτικού ελέγχου αποστεριόρι, εκ των υστέρων. Διότι η εγκύτητα, η ε, και η διαχείριση και η εκτέλεση των δράσεων δεν θα επιτρέπει μια απριόρι προηγούμενα εξάντε δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν ε, ε, εκ των υστέρων να διασφαλίζουμε εμείς αυτό τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία ε, τέθηκαν και τίθενται όσον αφορά την φύση των οργάνων αυτών και είναι μια άλλη πτυχή των προβλημάτων που πρέπει να επιλύσουμε. Επιμένω και εμένω, δεν ξέρω αν θα ήταν σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε κάπως τον ορίζοντα τον, ε, το πλαίσιο και την εμβέλεια, τον ορίζοντα αυτών των οργανισμών και θεσμών. Και αν υπάρχει μια τελική καθοριστική, ας το πω έτσι, ε, λύση για αυτά τα θέματα, να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία όσον αφορά την έκθεσή μας. Ευχαριστώ. Μέντες. Μέντες Πρόεδρε, Πρώτα, Εύνερ, παρακαλώ. Και θα ήθελα, λέει ο κύριος Μέντε Τεβίγο, αν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τη δική της άποψη, θα ήθελα να ακούσω την άποψή της. Ευχαριστώ. Κυρία Τάν είχε ζητήσει όμως τον λόγο πιο πριν, πριν από μένα. Ε? <laughs> Ναι, σας ευχαριστώ για αυτή την επισήμανση και αναφορά. Θέλω και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου στους δύο προλαλήσαντες και να πω ότι πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή και ας το πω υπό το γερμανικό πρίσμα μια ανεξάρτητη χρηματοεποπτική αρχή και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εγγυάται αυτή η αρχιτεκτονική. Οι διαφάνειες ήδη έδειξαν ότι τα θέματα αυτά είναι αρκετά περίπλοκα και λόγω της απουσίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εδώ υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορούν να προβλεφθούν ότι θα ε, δημιουργηθούν. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, διασφαλίζει πολύ μικρή ανεξαρτησία και εμείς στη Γερμανία με δύο αρχές επιτήρησης, μία ομοσπονδιακή και μία άλλη, είχαμε κακή πείρα, κακή εμπειρία και θα έπρεπε να υπάρχει μία ενιαία εποπτική αρχή. Και σε αυτή την αρχή δεν ανταποκρίνεται το σύστημα το οποίο μας παρουσιάστηκε. Γι' αυτό θα έπρεπε να δώσουμε συνέχεια στην πρόταση ή να αναμείνουμε λίγο παραπάνω για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά η λήψη απόφασης ή να υποβάλουμε δικές μας ξεχωριστές προτάσεις για να διασφαλιστεί αυτή η πτυχή και να προσπαθήσουμε, να το πω έτσι, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε στην Επιτροπή οικονομικό Οικονομικών Νομισματικών, να ασκήσουμε επιρροή ώστε να επιτευχθεί αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Βρισκόμαστε στην πολύ πρώτη στην ας το πω έτσι ψηλάφιση, ε, ας το πω έτσι ανείχνευση των θέσεων και των προβλημάτων. Αυτό είναι η ψηλάφιση ανείχνευση και σε αυτή την πρώτη φάση νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Μέντεθ Βίγο για το υλικό που δίνεται για τις περαιτέρω διαβουλεύσεις και περαιτέρω συνέχεια. Να ξεκινήσω διαφορετικά. Πιστεύω εγώ ότι εδώ για την ε, συγκρότηση αυτή μέσω των συνταγματικών θεμάτων θεωρούμε ότι δεν ήταν ίσως, ε, θεωρήθηκε ότι δεν θα ήταν ίσως αναγκαίο να διασφαλιστεί αυτή η πτυχή. Και έτσι τα θέματα αυτά δεν είναι καθόλου μόνο οικονομικού χαρακτήρα. Το κύριο ερώτημα που βρίσκεται στον πυρήνα όλων αυτών είναι πώς το νομικό πλαίσιο μπορεί να δημιουργηθεί για όλα αυτά που έχουν οικονομική συνιστόσα και πτυχή μέσα σε μια ελεύθερη οικονομία της αγοράς αλλά όμως προφανώς που δεν μπορούν να πετύχουν προ όφελο όλων αν λείπει αυτό το γενικότερο, ευρύτερο νομικό συνταγματικό πλαίσιο. Και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε πληθώρα οικονομικών θεμάτων, αλλά έχουμε και πληθώρα συνταγματικών και νομικών, νομικών θεμάτων. Είναι δύσκολο όλα αυτά να αποτιμηθούν σωστά και να υπάρξουν οι σωστές διαχωριστικές γραμμές υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να μας κάνουν να λάβουμε υπόψη και συνταγματικές πτυχές και την ανάγκη να έχουμε μια ενιαία έκθεση με έναν ενιαίο εισηγητή ώστε να είναι καρποφόρο το εγχείρημα και να είναι γόνιμο το εγχείρημα. Εκτιμώ και συμμερίζομαι την ε, εκτίμηση άλλων προλαλισσάντων ότι βρισκόμαστε στα σπάργανα ακόμα, στις απαρχές, στα πρώτα βήματα αυτή της εξέτασης και συζήτησης και θα ήταν λάθος να εγκρίναμε υπερβολικά βιαστικά μια πρόταση νομίζοντας ότι έτσι επιλύουμε όλα τα προβλήματα. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα από αυτό και χαίρομαι ότι και από διαφορετικές πλευρές αναφέρθηκε στη συζήτηση αυτό το στοιχείο και αναφέρθηκε ότι ιδιαίτερα εμείς ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από το σημερινό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Να έχουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες να ασκήσουμε επιρροή. Θέλω να αφήσω τα πράγματα σε αυτό το σημείο γιατί μπορούμε σε υστερότερη φάση να ξεκινήσουμε στην εμβάθυνση αυτών των θεμάτων. Αυτή είναι η προσανατολισμή για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί. Ευχαριστώ. Adesso και τώρα νομίζω πως δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν να πάρουν το λόγο. Η εκπρόσωπος λοιπόν της Επιτροπής θα πάρει το λόγο, κυρία Τσάισεν. Α, ο κύριος Τσάισεν. Ευχαριστώ πολύ, Τσάισεν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Αγορών. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων. Πιστεύω πως πολλά από τα ερωτήματα και πολλές από τις συζητήσει που κάνετε είναι παρόμοιε με αυτές που εμείς κάναμε όταν προετοιμάζαμε αυτή την πρόταση. Προσπαθούμε να βρούμε λύση για να κάνουμε μια πρόταση που να προτείνει ένα σύστημα το οποίο να είναι δυνατόν μέσα στο υπάρχον πλαίσιο, ισχύον μάλλον πλαίσιο τη συνθήκη τη Λισαβόνα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο όσο περισσότερο γίνεται να βρούμε φιλόδοξες και λειτουργικές λύσεις ώστε να βελτιωθεί η εποπτεία εντός της Ένωσης και νομίζω πως θα είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση η συζήτηση μαζί σας από αυτό Σίγουρα κάποιες από αυτές τεχνικές πτυχές σχετίζονται με νομικά θέματα, όπως για παράδειγμα σε ποιο βαθμό οι συνθήκες επιτρέπουν την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τέτοιου είδους οργανισμούς και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που σχετίζονται και με το θέμα του ρόλου της Κομισιόν Προσπαθούμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο προς την ανεξαρτησία, προς ανεξάρτητες ε, αρχές ε, που αποτελούνται από πυρογνώμονες, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι το πλαίσιο της συνθήκης απαιτεί ε, περιορισμού στο τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως ευχαρίστω θα σας πούμε οτιδήποτε άλλοτε οτιδήποτε άλλοτε χρειαστεί κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριο Μέντε να ολοκληρώσει. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας σε όλους τους προλαλήσαντες ότι τους ευχαριστώ για τα λόγια τους και τις παρεμβάσεις τους. Όπως είπα στην αρχή αυτή η ανταλλαγή είναι μια ανταλλαγή απόψεων. Είναι θετικό αυτό και ως ανταλλαγή απόψεων την αντιμετωπίζω. Έχοντας ακούσει όλους, βλέπω, και αυτό αναφέρθηκε, ότι το θέμα είναι ακόμα ανώριμο, δεν έχει οριμάσει ακόμα, είναι άγουρο και έτσι δεν έχει με κανένα τρόπο ολοκληρωθεί γιατί, διότι για πολλούς λόγους και για δύο λόγους που προαναφέρθηκαν πιο πριν και από τον κύριο Χάουρεγγι ε, και ότι εσείς κύριε Χάβνερ έχετε, έχετε δίκιο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Σεπτεμβρίου 2009 είναι μια αντίδραση στη χρηματοοικονομική κρίση. Εντάξει, μια αντίδραση σε αυτήν. Και αυτό επειδή αυτή η φιλοσοφία πολιτική φιλοσοφία και έμπνευση να μην υπάρξει παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αφήσουμε τα πράγματα στο κρατικό επίπεδο, δεν λειτουργήσε σωστά. Λοιπόν, αυτή είναι η αξιολόγηση. Δεν λειτουργήσαν τα πράγματα λοιπόν στο παρελθόν με την κρατική παρέμβαση. Τώρα πρέπει να γίνει κάτι καινούριο, σε ευρωπαϊκή παρέμβαση. Και είναι πολύ πιο δύσκολο λοιπόν να δει κανεί τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει και πώ μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να έχει νόημα και λόγο ύπαρξη και φυσικά η αντίδραση είναι πρέπει να έχει νόημα, εκείνο το οποίο συνέβη στο παρελθόν δεν πρέπει να επαναληφθεί, να επαναληφθεί χρηματοοικονομική κρίση και Τώρα, για τη δημιουργία θεσμικών οργάνων ή ε, υπηρεσιών ε, που μπορεί να μην έχουν σαφείς αρμοδιότητες ή να μην έχουν ένα σαφές πλαίσιο και ένα σαφή χαρακτήρα και να μην έχουν όλα αποσαφινιστεί επαρκώς. Είναι ένα θέμα λοιπόν πάρα πολύ περίπλοκο και καθόλου απλό, διότι επιπλέον δημιουργούμε, χτίζουμε σε μια σε παρθένα γη, σε άγνωστο ε, πεδίο και πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει νομική διαμόρφωση πραγμάτων για ε, την διαμόρφωση, ε, την σωστή αντιμετώπιση πολιτικών επιταγών και αναγκών. Δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει λοιπόν να ακολουθηθεί μια στρατηγική σωστή. Αναφέρθηκε αυτό και από τον κύριο Φεχόφστατ και από άλλους. Λοιπόν, τι είναι εκείνο το οποίο γίνεται και κάνουμε προχωράμε και προτείνουμε στην, Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ένα θεσμικό πλούς πλαίσιο για αυτές τις τρεις αρχές ε, και για το Συμβούλιο ε, ε, Συστημικών Κινδύνων. Μια δυνατότητα μπορεί να είναι αυτή. Ή θα αναμείνουμε να δούμε τι θα γίνει, τι γίνεται, τι, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αντίστοιχα θα αντιδράσουμε και θα τοποθετηθούμε. Και μήπως ε, ε, πρέπει να δούμε ότι υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί μικρότερη επιρροή από πλευράς μας. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος να προτείνουμε κάτι το οποίο θα απορρίψει στο τέλος τέλος ε, η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Λοιπόν, με τέσσερις διαφορετικούς εισηγητές ε, κιόλας επιπλέον, ε, εσείς έχετε εμένα ως ε, μόνο εισηγητή. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, αλλά με τέσσερις εισηγητές τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Λοιπόν, το θέμα για το νόημα της στρατηγικής, πολύ σωστά τέθηκε. Τι θα κάνουμε, τι πράγμα θα επιλέξουμε και πώς θα κινηθούμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποσαφηνίσουμε περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο με ανησυχεί πολύ αυτές τις στιγμές. Και αυτό ποιο είναι. Είναι ο συσχετισμός μας με την Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων. Διότι θα προχωρήσουν από πλευράς της Επιτροπής ΕΚΟΝ σε αυτό το θέμα. Θα έχουν ακρόαση και ε, αύριο και θα έχουν έγγραφα επιτραπέζης και στοιχεία και να μην ξεχνάμε και αυτό περιπλέκει τα πράγματα ακόμα παραπέρα ότι κάνουμε λόγο για συναπόφαση. Δεν αξίζει να κάνουμε κάποια γνωμοδότηση με κάποιες συστάσεις προς τη μία ή άλλη κατεύθυνση. Καθόλου πρέπει να πούμε, μια και κάνουμε λόγο εδώ, γίνεται λόγος για technical standards και έχουμε εδώ μια πρόταση της Επιτροπής και υπάρχουν προτάσεις του Συμβουλίου, εμείς ως Ευρωβουλή πρέπει να διατυπώσουμε εναλλακτικές προτάσεις. Πρέπει νομικά να τις διατυπώσουμε με επαρκή τρόπο, με επαρκή μορφή και πρέπει να πω απλά ότι το θέμα αυτό δεν είναι καθόλου απλό και καθόλου εύκολο. Κύριε Φερχόφστατ, για την ικανότητά σας ε, να ε, θέλγετε το ε, ισπανικό σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και τον κύριο Θαπατέρο που γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμω, κύριε Φερχόφστατε επιτρέψτε μου αυτό το αστείο. Εντάξει. Εσείς τι μα προτείνετε κύριε Φερχόφστατε. Να αλλάξουμε πλήρω πρότυπο. Και λέτε γιατί τρει αρχέ, Όχι μόνο μία ενιαία αρχή και έτσι λοιπόν να μπορέσουμε να ναι. ε, προχωρήσουμε καλύτερα. Εδώ θα πρέπει να αναζητηθεί συνένεση. Αυτό θα σημαίνει ρήξη όμω ε, με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το Συμβούλιο συμφωνεί επ' Πρέπει να έχουμε πολλά λοιπόν επιχειρήματα πολιτικά, νομικά, οικονομικά για να μπορούμε να προασπίσουμε μια τέτοια θέση. Και όταν κάνουμε λόγο για συναπόφαση, και εδώ έχουμε μια αρχή που όλοι συμμεριζόμαστε, που είναι το μονοπόλιο στην άσκηση πολιτική πρωτοβουλία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει αυτό να το δούμε και να διαφυλαχθεί σε ένα τόσο θεμελιώδες ε, σημείο. Και αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Τούτων λεχθέντων, κύριε Σμιτ, σα ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σα. πιστεύω ότι οι τρεις αρχές ε, εποπτείας ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εκείνο που δεν έχει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι η Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων. Οι άλλες έχουν. Είπατε κάτι και είναι ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι η ιδέα της θέσπισης ε, προθεσμιών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στην επίλυση ε, τριβών ή προβλημάτων που μπορούν να δημιουργούνται ή όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, πρέπει να θεσπίζονται πρώτο, με προθεσμίες. Δεν μπορούν να αφήνονται τα πράγματα χωρίς άλλη ρύθμιση μέσα σε ένα ανοιχτό πλαίσιο. Αυτό έχει σημασία, έχει ρόλο κλειδιού. Και εδώ στο τέλος τέλος για την πρόταση της Επιτροπής όταν δεν υπάρχει συμφωνία, λέει, θα λαμβάνει απόφαση και θα ρυθμίζει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκείνο που πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά είναι η νομική φύση των πράξεων των ε, Ευρωπαϊκών Αρχών ε, Εποπτείας. Η σχέση τους ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιου, λόγου, για ποιου είδους πράξεις και παρεμβάσεις κάνουμε λόγο. Και εδώ για, δεν κάνουμε λόγο μόνο για την εκ των υστέρων δυνατότητα ελέγχου. Κάνουμε λόγο για την δυνατότητα δράσεων που μπορούν να υποστηριχθούν αποστεριόρι ή να εγκριθούν ή και όχι θα, θα πρέπει να δούμε ότι θα είναι πάρα πολύ περίπλοκο να ενταχθεί η πρόταση αυτή σε σχέση με αυτό που πρέπει να γίνει, το είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στο πλαίσιο της συνθήκης. Είμαστε μια κοινότητα δικαίου και όταν κάνουμε πράγματα όσον αφορά την, ε, τον πιο ενδεδειγμένο χαρακτήρα που μπορεί να έχουν ή τον πιο σκόπιμο ρόλο που μπορούν να έχουν, εκείνο που αποτελεί κριτήριο είναι το πλαίσιο των συνθήκων, οι κανόνες του παιχνιδιού που δεν μπορούν να αλλάζουν και να αλλοιώνονται. Και ο δεσμευτικός ε, ε, λόγος, ο δεσμευτικός ρόλος τέτοιου είδους συστάσεων ή παρεμβάσεων και να δούμε πώς θα παρεμβαίνει στο τέλος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ολοκληρώνοντας, Πρόεδρε, σημειώνω όλα τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοι Αύριο θα παραστώ στην, Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων και θα δω ποια κατεύθυνση ακολουθούν οι εισηγητέ αυτή τη Επιτροπή, τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Και πιθανότατα πιστεύω ότι θα χρειαστούμε και άλλη συνεδρίασή μα για να εμβαθύνουμε σε αυτά τα θέματα και μετά από αυτήν θα έχοντας ε, ε, σκεφτεί σε βάθος και έχοντας δει προς τα που θα κινηθεί η Επιτροπή Νομισματικών ε, Οικονομικών να δούμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φερχόφστατ να έχουμε φιλόδοξο πλαίσιο στις δράσεις μας και να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η φιλοδοξία από πλευράς μας και να δούμε σε σχέση με την τοποθέτηση την αρχική όσον αφορά την τοποθέτηση της ΕΚΟΝ η δική μας δεν ήταν επαρκώς φιλόδοξη να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πιο φιλόδοξη πρόταση. Θα έρθω σε επαφή με τους τέσσερις εισηγητές, θα ε, δω πού βρισκόμαστε και αυτό θα μου δώσει τη δυνατότητα να είμαι καλύτερα πληροφορημένος και να σας διαβιβάσω πού βρισκόμαστε και πώς κινούμαστε σε αυτή την σε εξέλιξη δραστηριότητα αυτής της αρχιτεκτονικής. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας για τις παρεμβάσεις σας. Parce que je voulais en fait σας ευχαριστώ. Ήθελα ακριβώς να προτείνω το ίδιο με αυτό που συμπέρανε στο τέλος ο κύριος Δεμέντες Δεβίγκο, να γίνει μια συνεδρίαση ανάμεσα στους τέσσερις συζητητές και τον ίδιο για να δούμε πώς εμείς στην Επιτροπή μας μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί βοηθούμε στη δουλειά τους για να είμαστε βέβαιοι ότι από θεσμική άποψη θα προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν πως αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ο μόνος λόγος ε, της δικής μου παρέμβασης, ε, κύριε Μέντες Δεβίγκο, είναι ότι θα υπάρχει μια συνδιαλλαγή ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για αυτή την υπόθεση. Αυτό μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Είναι συναπόφαση, δεν έχουμε ακριβώς την ίδια θέση. Ε, πιστεύω πως ακόμα και από την άποψη της ε, Ισπανικής Προεδρίας υπάρχει μια θετική θέση απέναντι σε προτάσεις που προχωρούν πιο μακριά. Το συζήτησα με την κυρία Σαλγάδο όταν κάναμε τη συνεδρίασή μας στη Μαδρίτη. Αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο και το μόνο πράγμα για το οποίο έχω παρέμβει είναι ότι η δική μας Επιτροπή και εσείς είστε θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε εκεί όπου βλέπουμε ότι οι, τρεις, οι τέσσερις ηγητές θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο να τους βοηθήσουμε. Γιατί στη συνδιαλλαγή θα χρειαστεί να δείξουμε ενότητα από πλευρά του Κοινοβουλίου γιατί διαφορετικά δεν θα πετύχουμε τίποτα. Και επιπλέον έχουμε τώρα και την ε, κλίση του κ. Μπαρόζο που λέει πρέπει να βοηθήσετε, πρέπει να βοηθήσετε. Γιατί η ΕΚΟΦΗΝ ε, θάβει, θάβει, σαμποτάρει τις προτάσεις μου. Ε, να το κάνουμε. Να προχωρήσουμε ακόμα λίγο πιο μακριά. Είμαστε κοντά. Ε, στη, είμαστε κοντά, λίγη κοινή λογική. Είμαστε κοντά, στο, όχι στο ιδανικό γιατί αυτό είναι ανύπαρκτο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα που μπορούμε να λειτουργήσουν καλύτερα από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Αυτό, αυτό το νόημα έχει η παρέμβασή μου. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Αυτή η υπόθεση τελικά είναι περίπλοκη μαζί με τις άλλες θα είναι έντονη η επόμενη περίοδο. Στην πράξη, οι πληροφορίε που έχουμε, δεν ξέρω αν ο Μέντε Δεβίκο έχει διαφορετικέ πληροφορίε, πάντως η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή θα ήθελε να ολοκληρώσει την εργασία τη τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν, αν εμεί θέλουμε να γνωμοδοτήσουμε, παρότι θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο να το σκεφτούμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο τελικά στη διάθεσή μα. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ένα έγγραφο Προσυζήτηση στις 22 Φεβρουαρίου. Είναι δυνατόν? Μάλιστα. 22 Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε. Όλα είναι δυνατά, αγαπητέ Πρόεδρε. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να ορίσουμε την επόμενη συνάντηση ή προσυζήτηση της 22 Φεβρουαρίου, ώστε να το εγκρίνουμε στις 7 Απριλίου. Αυτό θα είναι το χρονοδιάγραμμα. Έχω την εντύπωση ότι εξαντλήσαμε όλα μας τα θέματα εδώ. Θα πρέπει μόνο να θυμίσουμε τις ημερομηνίες των προσεχών μας συνεδριάσεων. Να θυμίσω ότι 8 Φεβρουαρίου θα είναι παρόν στο Στρασβούργο ο ε, Υπουργό Εσωτερικών Λόπε Γκαρίδο. Στι 22 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη μα συνεδρίαση τακτική στι Βρυξέλλε. Το πρόγραμμα προέβλεπε και συνάντηση των συντονιστών. Μπορούμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί να, για τις 6.30 οι διερμηνείς θα φύγουν. Έχουμε ένα τεταρτάκι. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε ένα τεταρτάκι και αν δεν τα καταφέρουμε θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια άλλη ευκαιρία για να τα πούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής. Παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν.